Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημέρα διάταξη. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις. Να υπενθυμίσω απλώς ότι έχουμε εγκρίνει δύο ψηφίσματα ε, επιγόντω μετά την Ολομέλεια του Ιανουαρίου η κατάσταση, η επίκουσα κατάσταση στο Μπουρούντι και ιδιαίτερα το θέμα της ελευθερίας έκφρασης και η κατάσταση στην Ιγυρία επίσης ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις. Δύο χώρες ε, της Αφρικής ε, που αποτελούν προτεραιότητα όπως αντιλαμβάνεστε Επίσης, την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο έκρινε την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Είναι η ετήσια έκθεση του 2018. Θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ την Ιζαμπέλ που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή αλλά και όλους τους συνεισηγητές για το έργο τους. Τρίτο σημείο, έγκριση των πρακτικών Έχουμε τα πρακτικά 11 και 12 Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Πολύ ωραία τέταρτο σημείο. Σήμερα ξεκινούμε το έτος 2020 με την ανταλλαγή απόψεων με τον Ήμον Γκίλμορ. Θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον Ήμον. Έχετε 10 με 15 λεπτά για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας στην αρχή των εργασιών σας για το 2020. Είχα έρθει στην Επιτροπή αυτή 9 Σεπτεμβρίου τελευταία φορά. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας ενημερώσω για κάποια από τα κεντρικά ε, σημεία των εργασιών μου έκτοτε και να σας πω βεβαίως και ποια είναι τα σχέδιά μου για το μέλλον, να ακούσω και τις δικές σας ανησυχίες, τις προτεραιότητες τις δικές σας. Όπως ξέρετε η απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου, 28 ε, Φεβρουαρίου, έρθει να προσθέσει στην εντολή ε, του εκπροσώπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων την, το καθήκον του να συνεισφέρει ε, στην βελτίωση, στην ενίσχυση του, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της διεθνούς ποινικούς, ε, ποινικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έτσι λοιπόν επισκέφθηκα τη Χάγη δύο φορές για να συναντήσω τις, ε, τους διεθνούς οργανισμούς που βρίσκονται εκεί και να εκφράσω βεβαίως την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το ποινικό δικαστήριο τον, στα μέσα Σεπτεμβρίου μαζί με τον κύριο Λέφλερ συνάντησα τον πρόεδρο και τον ε, κεφαλής, τον, τον εισαγγελέα της ε, ε, ICC, τους υπεύθυνους για την υπόθεση του Κωσυφοπεδίου, ήταν εγκλήματα πολέμου εκεί, επίσης τον υπεύθυνο για τους αγνοούμενους και τον αντιπρόεδρο του Eurojust, τον γενικό διευθυντή της οργάνωσης για την απαγόρευση των χημικών όπλων. Συνάντησα επίσης ε, στο, στις Βρυξέλλες στον εκπρόσωπο ε, της, του δικαστηρίου για το Κωσυφοπαίδιο ε, έγινε και μια εκδήλωση τον Δεκέμβριο που ε, Φιλανδικής Προεδρίας για την υποστήριξη της ICC είναι σημαντικό ε, να υπάρξει συμμόρφωση με την ICHO και την ICJ και να υποστηρίξουμε το έργο της ICC. Εγώ υποστηρίζω την απόφαση του Μπάτη ε, να επικυρώσει, αλλά παραμένουν ακόμα ε, αρκετές χώρες ε, που δεν έχουν επικυρώσει το, το, τη σύμβαση για το ICC. Κάποιες χώρες επίσης που είχαν ζητήσει να αποσυρθούν το ξανασκέφτονται, αυτό είναι θετικό. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες επίσης συμπροέδρευσα την, το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αφρικανική Ένωση, τη Βραζιλία, την Κούβα, ε, την Νότια Αφρική ε, και είπα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια. Αυτός ο διάλογος δηλαδή δεν πρέπει να είναι απομονωμένος, να αποτελεί μέρος, πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας με τις εν λόγω χώρες ή με τις εν λόγω ε, περιφερειακές οργανώσεις για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση της Αφρικανικής Ένωσης συμφωνήσαμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες για την μεταβατική δικαιοσύνη ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. την Νότια Αφρική ενθαρρύναμε την συμμετοχή ε, στην ε, πρωτοβουλία για, τα, για τις καλές ιστορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τις ονομάζουμε. Με την Κούβα συμφωνήσαμε ότι υπάρχει περιθώριο για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας για την προστασία των δεδομένων και για την, βία, την έμφυλη βία και για την περίπτωση της Βραζιλίας η βραζιλιανική πλευρά μας προσκάλεσε να επισκεφθούμε το, τη χώρα αυτή πριν το επόμενο διάλογο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα ζητήματα που συζητήσαμε το φθινόπωρο. Πέρα από τους διαλόγους αυτούς, οργανώσαμε για πρώτη φορά από το 2015 διαβουλεύσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις ΗΠΑ ε, Από την Αμερικανική πλευρά συμμετείχε ο νέος υφυπουργό ε, εξωτερικών για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασίας, ο κ. Ρόμπερτ Ντέστρο. Η συνεδρίαση αυτή ήταν σημαντική όχι μόνο επειδή ήταν η πρώτη μετά από τέσσερα χρόνια αλλά και διότι ε, έχετε μετά την ε, απόσυρση των ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βεβαίω υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα όπως η δημιουργία μιας επιτροπής ε, για τα αναφέρετα δικαιώματα. Είχαμε και μια συνάντηση στη Washington και στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2019 και αυτό η συνάντηση ήρθε ως συνέχεια, ως συνέχεια. Θα επισκεφτώ τη Washington για περαιτέρω συζητήσεις τον ερχόμενο μήνα. Αποκινούμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με την Αφρικανική Ένωση. Τον Οκτώβριο επισκέφτηκα την Γκάμπια. Εκεί είχαμε πολύ σημαντικέ αλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσει μια διαδικασία ε, για ένα νέο σύνταγμα που αποτέλεσε αντικείμενο μια καινοτόμας Διαδικασία δημόσια διαβούλευση. Ε, δίνει τη μεγάλη έμφαση εκεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθεί ε, να ηγηθεί στα ζητήματα αυτά στο μέλλον ε, τουλάχιστον αυτό που δείχνει και η δράση η νομική χαρά της Μιαμάρ ήμουν και στην τρίτη πρωτοβουλία προέδρευσα την τρίτη πρωτοβουλία για τις καλές ιστορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νότια Αφρική το τέλος του λόγου μίσους κατά τον ε, ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, η προστασία της θρησκευτική ελευθερίας, το πάνελ για την επανοικοδόμηση των κοινοτήτων και των ζωών ε, και η ομάδα φίλων της Συμμαχίας των Πολιτισμών. Υπάρχει και εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων των ε, επιζώντων σεξουαλικής βίας. Συνάντησα τη Μισελ Μπασλέ, συνάντησα ε, τον Πίτρε Μέρερ από την ICRC, και ε, τη Βιτζίνια Γκάμπα που ασχολείται με τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες. Είχα και δημιουργήσει επαφές ε, για να δώσουμε συνέχεια στις νωρίτερες συζητήσεις, στις ε, συναντήσεις του 2019, συνάντησα την Υπουργό Εξωτερικών της Μιαμάρ, του Μπαγκλαντές και της Ερυθρέας. Επίσης είχα μια συνάντηση με τον ειδικό εκπρόσωπο, την ειδική εκπρόσωπο την Κρίστιαν Μπέργκελερ, των ΗΠΑ στη Μιαμάρ με τη Λευκορωσία συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Βλαντιμίρ Μακέη. Επίση συνάντησα τον νέο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, ε, τη Μαρία Πετσένοβιτ Γκούριτ και ε, τον εκπρόσωπο ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συνάντηση στην επίσκεψή μου στο Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο όπου έγινε η παρουσίαση του βραβείου Ζαχάροφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την ε, τελετή αυτή συνάντησα ξεχωριστά την Τζούλεν Χάλχαμ που έλαβε ε, το ε, βραβείο στο όνομα του πατέρα της ε, και συνάντησα βεβαίως και τον ακτιβιστή από τη Βραζιλία και τις, τα από την Κένια που έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο για την προστασία των κορίτσων και των γυναικών εκεί. Ήταν οι δύο άλλοι υποψήφοι. Επίσης ήμουν ε, στο Ευρωπαϊκό Μάστερ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στην Βενετία τον Οκτώβριο σχετική τελετή ε, αποφύτησης ε, το Δεκέμβριο ε, πήγα στη Βιέννη στην Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων για να εξετάσω πόσο αυτή η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έρευνα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων, πώ μπορεί να συνεργαστεί με το δικό μου γραφείο και με την, Ευρωπαϊκή, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών τη Ένωση και των εξωτερική και εξωτερική δράση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το Σεπτέμβριο μίλησα σε πολλέ διασκέψει και εκδηλώσει για να προωθήσω το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα σχετικά θεσμικά όργανα για τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Ε, μίλησα επίση στην ε, Ένωση ε, Δικαστικών και Εισαγγελέων για το κράτο δικαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην, στο φόρουμ το ΜΚΟ όπου η HRVP ε, ε, έκανε την πρώτη της ομιλία για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το που τη θητεία τη. Ε, συνάντησα πολλέ συναντήσει κοινωνία των πολιτών, πολλέ οργανώσει κοινωνία των πολιτών για πολλά και διάφορα ζητήματα, καθώ και εκπροσώπου για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαφόρων εθνικών χωρών. Θα πάω στη Λευκορωσία μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη. Με έχουν προσκαλέσει και στην Ουκρανία. Ο Δημήτρη Κολύμπα, ο αντιπρόεδρο με συνάντησε πρόσφατα για το ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες. Πρόκειται να, να επισκεφτώ και το Μεξικό για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για διμερή, ενδεχόμενη διμερή συνάντηση. Ελπίζουμε αυτό να γίνει στην αρχή του 2020 μετά την επίσκεψη τη Υπηρεσία Ανθρωπίνων τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κατάρ με κάλεσαν σε μια διάσκεψη μέσα Φεβρουαρίου στην Τόχα. Ε, Εξέφρασε το ενδιαφέρον να επισκεφθώ την Αίγυπτο. Συνάντησα και τον πρέσβη τη Αιγύπτου για το ζήτημα αυτό. Ο, πρόσφα... πρέσβη του Πακιστάν με συνάντησε πρόσφατα. Ενδεχομένω να επισκεφθώ λοιπόν και το Πακιστάν αργότερα φέτο. Ε, ενδεχομένως ταυτόχρονα με την επόμενη συνάντηση της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης που θα λάβει η χώρα στο Πακιστάν. Έχει, σκεφτόμαστε επίσης να έχουμε επαφές με τη Σαουδική Αραβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο με, καν, με κανόνες που δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτοί από, τους, από τη Σαουδική Αραβία όταν επισκέφθηκε το εκπρόσωπο τη Τουρκία Αυγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι Βρυξέλλε τον συνάντησα τον Δεκέμβριο και συνάντησα και τον κύριο Αλτζαμπίρ πολύ πρόσφατα. Με ήρθα σε αυτή την επιτροπή, επισκέφθηκα το Σεπτέμβριο ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περαιτέρω συζητήσει μαζί σα, κυρία Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη επίση ενημερώνονται για τι εργασίε μου. Ε, πήγα λοιπόν στην PSC μετά την τελευταία συνάντησή μου και έδωσα σχετική αναφορά και ήμουν και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 9 Δεκεμβρίου. Όπω ξέρετε, έγινε εκεί μια ειδική συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα αποτελέσματα αυτή τη συζήτηση, καθώ και η περαιτέρω σκέψεις ε, για το σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία θα ε, με απασχολήσουν σημαντικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτέ είναι ε, και άλλε πολλέ είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στα ζήματα των δικαιωμάτων, πολλές, σε πολλέ χώρε και περιφέρειες του κόσμου, κάτι που μα υποχρεώνει να συνεργαζόμαστε ακόμα πιο στενά. Είναι πολύ σημαντικό το έργο τη Επιτροπή αυτή και αναμένω σήμερα να ακούσω τις σκέψεις σας, τις σα, τι προτεραιότητέ σα και να έχουμε άλλη, άλλον ένα επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα τους ομιλητές, η Ιζαμπέλ Σάντος πρώτη. Η Ρίνα, Άννα, Χάιντι. Δίνω το λόγο στην Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Βάλτε τα ακουστικά σας, λοιπόν. Καταρχήν θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2020. Ξεκινήσατε το έργο σας περίπου ένα χρόνο νωρίτερα για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια εποχή που η κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και είχαμε μια πολύ καλή παρουσίαση για την κατάσταση στις διάφορες χώρες, ε, το διάλογο. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Θα ήθελα όμως ε, να το δούμε αναχώρα και να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Για να δούμε και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Έχουμε κάνει, έχουν γίνει διμερείς συνομιλίες με τη Βραζιλία. Ο Ιθαγιανής πληθυσμός εκεί ζει σε συνθήκες που δεν ξέρω αν συζητήθηκαν στις ομιλίες σας. Ο λόγος μίσους κατά της κοινότητας των LGBT συζητήθηκε στις συζητήσεις σας. Η χρήση βίας έως θανάτου από την οικονομία, από την αστυνομία, συγγνώμη. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που προέκυψαν πρόσφατα, αποκαλύπτεται ότι πεθαίνουν κάθε μέρα 17 άτομα στα χέρια της αστυνομίας. Συζητήθηκε κάτι τέτοιο ή είναι μεταξύ των θεμάτων που θέλετε να συζητήσετε στο μέλλον όσον αφορά την Κούβα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν το φύλλο, την προστασία δεδομένων και θα ήθελα να ρωτήσω αν συζητήθηκε και το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Το θίξατε αυτό το θέμα. Για τις Ηνωμένε Πολιτείες μιλήσατε και εκεί με τους ομολόγους σας. Είχαμε και εμείς μια αποστολή στις Ηνωμένε Πολιτείες και είχαμε συζητήσεις και μιλήσαμε με τον κύριο Ντέστρο κατά την αποστολή αυτή. Για τις Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, η δημιουργία μιας ε, Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι αξιέπαινη προσπάθεια και πολύ σημαντική ε, προέκυψε το θέμα των, ε, του μεταναστευτικού ιδίω των μεταναστών από τη Λατινική Αμερική που προσπαθούν να μπουν στις Ηνωμένε Πολιτείε και το τι γίνεται με τους μετανάστες αυτούς ιδίως όταν αποκόπτονται από την οικογένειά τους προέκυψε το θέμα της θανατικής ποινή. γιατί είναι μια συζήτηση που έχει γίνει ε, αρκετά τελευταία σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινή σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Συζητήθηκε στις ε, συνομιλίες σας. Επίσης, θα θέλετε να μας πείτε και τι προτίθεστε να συζητήσετε στο μέλλον για τη Σαουδική Αραβία μετά από όσα έγιναν χτες. Σας εύχομαι καλή τύχη στο διάλογο αυτό γιατί είναι τεράστια η πρόκληση. Και ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία γιατί χθες μου δόθηκε η εντύπωση ότι ο διάλογος αυτός δεν λειτουργεί καθόλου. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω ότι εσείς θα τα καταφέρετε θαυμάσια όταν θα συζητήσετε με τη Σαουδική Αραβία. Σχετικά με τη Λευκορωσία. Και εκεί υπάρχει το θέμα ε, της ε, θανατικής ποινή. Είναι ένα από τα θέματα που θέλετε να συζητήσετε με τη Λευκορωσία. Αυτά είχα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στην Ιρένα. Ειρήνα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκίλμο. Ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση για το διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και πιο συγκεκριμένα, εάν πιστεύετε ότι μετά την αποχωρήση ε, των Ηνωμένων Πολιτειών από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν ε, βλέπετε μεγαλύτερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιο είναι το μέλλον της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολυμερείς συζητήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, υπάρχει προοπτική να ξαναμπούν στο Συμβούλιο και τι, σημαίνει, ε, τι σημαίνουν όλα αυτά για την συνεργασία στο μέλλον. Επίσης, παρατήρησα ότι έλειπε μία χώρα από τον εντυπωσιακό κατάλογο που μας αναφέρατε για τους διαλόγους, η Ινδία. Έχετε κάνει καθόλου συζητήσεις με την κυβέρνηση της Ινδίας. Θα προσθέσετε την Ινδία στο κατάλογο των χωρών με τις οποίες συνομιλείτε. Αναφέρετε μια πιθανή επίσκεψη στο Πακιστάν. Νομίζω ότι θα ήταν λογικό να συμπεριληφθεί και η Ινδία στο πλαίσιο αυτό για να αντιμετωπιστεί η κρίση σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εκ μέρου των Πρασίνων, Άννα. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε κύριε Γκυλμό για την επίσκεψή σας. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πρόγραμμα που μας παραθέσατε από τους τελευταίους έξι μήνες δεδομένου ότι έχετε ε, τώρα κλείσει περίπου ένα χρόνο σε αυτή τη θέση και έχετε κάνει και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές συνομιλίες, η ερώτησή μου είναι τι έχετε προσδιορίσει ως βασικές θεματικές προτεραιότητες για τη θητεία σας στο μέλλον. Και δύο πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, πρώτον, αναφέρατε το διάλογο με τη, Βραζι... με τη Βραζιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι είμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευση Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Βραζιλία, θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη. Σε τι βαθμό πιστεύετε από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι πρέπει να συνεχίσουμε ή να αναστείλουμε ή και να διακόψουμε αυτέ τι συνομιλίε και με βάση τις συζητήσεις που είχατε για τη Μερκοσούρ. Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ε, για το διάλογο με τη Σαουδική Αραβία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μία επιπλέον ερώτηση. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το καθεστώς κυρώσεων εδώ και αρκετό καιρό και τώρα ε, θα θέλαμε ε, να ακούσουμε και τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε τη θέση σας επ' αυτού. Και για μελλοντικές συζητήσεις που θα κάνουμε μαζί σας, θα μπορούσατε να μας, δώσετε, να μας δίνετε εκ των προτέρων ε, τον προγραμματισμό των συνομιλιών σας ή να δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας ώστε να προγραμματίζουμε καλύτερα τις συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Φιλ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ξεκινήσω με το Πακιστάν και την επίσκεψη στο Πακιστάν. Εγώ είμαι σε συνεχή συζήτηση με την κυβέρνηση του Πακιστάν σε μεγάλο βαθμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική κατάσταση σε σχέση με το Κασμίρ. Θα μιλήσετε με τον κύριο Καρέσι όταν θα πάτε στο Ισλαμαμπάντ. Θα μιλήσετε για την γενική κατάσταση στο Κασμίρ είναι ένα από τα θέματα της μερικής διάταξης. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο να έρθω, γιατί έπρεπε να ψηφίσω το ψήφισμα για την Ινδία, που είναι στην άλλη άκρη του, του κτηρίου και επειδή υπήρχε κάποια προθεσμία, έχασα την αρχή της παρουσίασής σας και σας ζητώ συγγνώμη. Ένα δεύτερο σημείο τώρα, σχετικά με την πιθανότητα συνομιλίας με τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι τώρα η θανατική ποινή ε, ξεπερνάει και το Ιράν. Τα, τα θύματα των, της θανατικής ποινής σιγά σιγά στη Σαουδική Αραβία πάνε να ξεπεράσουν το Ιράν που είναι πρωταθλητή σε αυτό το κομμάτι. Επίσης για τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη. Μπορεί να συνομιλήσετε με τους Σαουδάραβες ε, ιδίως για την νότια Ιεμένη, γιατί κατά καιρού ακούμε ε, για ε, ελλείψεις ειδών διατροφής στο AIDEN και από την εκλογική περιφέρεια από το ε, ακούμε πολλά σχόλια για τις αποστολές τροφίμων και ανησυχούν πολύ για την αποστολή τροφίμων στο AIDEN όπου υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Αν και εμείς βγαίνοντα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μικρότερη συμμετοχή πλέον. Ευχαριστώ πολύ, Ιζαμπέλα. Ζητώ και εγώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι εδώ στην αρχή της παρουσίασής σας. Ζητώ συγγνώμη, παρότι θα ήθελα, δεν τα κατάφερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της κατάστασης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η έκθεσή σας και τα σχετικά έγγραφα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα του Βιετνάμ Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε την συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συμφωνία και θα θέλαμε τη δική σας άποψη. Από ό,τι βλέπω, σε κάποιους τομείς υπάρχει βελτίωση, σε άλλους δεν υπάρχει και τόση βελτίωση. Γι' αυτό θα ήθελα τη δική σας άποψη. Ακόμη θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη δική σας εικόνα σχετικά με το διάλογο μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης στη Βενεζουέλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλ, Χάιντι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον ειδικό εντεταλμένο που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας και μας έκανε αυτή την πληρέστατη παρουσίαση. Επανέρχομαι σε κάποια από τα σημεία που αναφέρατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που μας είπατε ότι στο διάλογο με την Αφρικανική Ένωση έγιναν συζητήσεις ε, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τομέα με τεράστιο ενδιαφέρον, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει στις εμπορικές μας συμφωνίες να βάζουμε τα θέματα επιχειρηματικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πώς θα διεξαχθούν οι συζητήσεις με την Αφρικανική Ένωση. Μιλάμε για τη σημαντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση και με όλες τις χώρες της Αφρικανικής Υπήρου και γενικά σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντική η χρονική στιγμή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται τις διάφορες προτάσεις που υπάρχουν για τη δέουσα επιμέλεια. Εσείς συμμετέχετε ενεργά σε αυτές τις συζητήσεις και μπορείτε να πείσετε την Επιτροπή να ακολουθήσει κάποια δράση, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται και μερικές επιτροπές μάλιστα με, μεγάλη, με μεγάλο ζήλο. Συνεχίζοντας σε αυτά που είπε η συνάδελφος η Χάνα Νόημαν, θέλω να πω ότι ότι το θέμα των κυρώσεων ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείστε με τις λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος, πώς θα γίνεται ακριβώς στην πράξη, γιατί θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση με, βάση τις δικές μας αξίες και τη δική μας κατανόηση του διεθνούς δικαίου και, τα, ε, ε, και του κράτους δικαίου. Τα διεθνή μοντέλα δεν είναι επαρκή και πρέπει να έχουμε τη δική μας προοπτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και να εκτραπεί προς κατευθύνσεις που δεν θέλουμε. Τέλος, μιλήσατε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου ζητούμε να υπάρξει μεγάλη δραστηριότητα σε αυτό το τομέα. Σε σχέση με την Παλαιστίνη είχαμε απρόσμενες εξελίξεις. Ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι, ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες. Ευχαριστούμε. Μπετίνα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, στα οποία υπάρχει απάντηση στην έκθεσή σας και θα ήθελα να περιστώ σε ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δεν αναφέρθηκε σήμερα. Στο πρόγραμμα εργασία σα θα συμπεριλάβετε και τον τομέα της δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίω, γιατί είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μεγάλο βαθμό και θα ήθελα να μας πείτε εάν έχετε την πρόθεση να ασχοληθείτε με το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Τέινα. Ευχαριστούμε κύριε Γκίλμορ Να σας το πω στα ισπανικά. Ονομάζομαι Ρίβα και είμαι πράσινη ευρωβουλευτής και έχω συνεργαστεί με τον κύριο Ρωμέβα, ο οποίος τώρα είναι πολιτικός κρατούμενος Καταλανός και το 2020 είχαμε, ε, έχουμε να αναλύσουμε τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε όλα και περισσότερες ε, παραβιάσεις δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ε, δύο με τρία δύο σταθμά. Αγνοούμε αυτά που γίνονται μέσα, στην Ένωση και είμαστε πιο κατηγορηματικοί αυτά που γίνονται έξω, πιο απόλυτοι. Οπότε θα πρέπει να έχουν περισσότερη συνέπεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, για πέστε μας ε, ε, σε αυτό το πνεύμα, ε, εσείς που είσαστε εκπρόσωπός μας, δεν θα πρέπει όλοι να συμμορφώνονται με τον χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Merci. Euh, je vais poser, poser une Έχω και εγώ μία ερώτηση, λέει η κυρία Αρένα, αν επιτρέπετε δύο. Σε σχέση με αυτό που είπαμε χθες στην Άφετ, ήρθε ο ΙΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας και δεν θα επανέλθω. Πώς απάντησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μου φάνηκε λίγο κλειστός αλλά η απάντησή του με προβλημάτισε τα δικαιώματα. Είπε ότι εσείς δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανέφερε το θέμα των μεταναστών και των δικαιωμάτων τους. Αλλά αυτό το πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τι κάνουμε και πώς ε, αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ένωσης. Οπότε, στο διάλογο αυτόν εσείς τι λέτε. Πώς το βλέπετε αυτό όσον αφορά το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπε ο Σαουδάραβας υπουργό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με τον διάλογο με τις σχετικές χώρες. Δεν θα πρέπει πρώτα να φροντίζουμε τα του οίκου μας πριν γινόμαστε κατήγοροι σε όλο τον κόσμο. Ένα αυτό. Δεύτερον, η υποεπιτροπή μας έχει προσπαθήσει, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους εισηγητές, ε, για το θέμα της συμφωνίας της εμπορικής με το Βιετνάμ και είχαμε ένα ενδιαφέρον ψήφισμα για το τι περιμένουμε από τη χώρα ως εμπορικό εταίρο. και δεν κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις σας. Οι συστάσεις μας. Οπότε, εσείς όπως είναι σήμερα τα πράγματα, πώς το βλέπετε. Για το Βιετνάμ θεωρείτε ότι είναι σε καλό δρόμο η χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν συναυθεί αυτή η συμφωνία, αν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τι κάνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να έχουμε ε, κάποια μέσα για να φροντίσουμε, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σας παραπέμπω και στην Βραζιλία, που και εκεί υπήρχαν διάφορες συμφωνίες, σύνδεσης, συνεργασίες. Όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό δεν είναι ένα θέμα αποστασιοποιημένο θα πρέπει να εντάσσεται στις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης με συνέπεια. Εσείς πώς το βλέπετε όσον αφορά τη συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συστάσεις σας. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Γκίλμουρ. Uh, for... Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Γκίλμουρ, για τις ερωτήσεις σας. Να απαντήσω. Πρώτα-πρώτα με την Βραζιλία. Προτεραιότητα για μένα και τα θέματα που ανέφερε η Ισαβέλ για τους Ινθαγενείς ε, και τα προβλήματά τους αυτά θα με απασχολούσαν όσον αφορά και τους ε, ακτιβιστές από αυτούς τη ρητορική μίσους κατά τον ΛΟΑΤΚΙ και κατά των γυναικών. Πολλά από αυτά έχω διαπιστώσει. Επίσης ότι γίνεται με την καταστολή των διαμαρτυριών και διαδηλώσεων και ήδη τα έχουμε συζητήσει στις επαφές με την χώρα. Όλα αυτά τα έχω συζητήσει και με ακτιβιστές βραζιλιάνους στην Frontline Conference και επίσης και με τον πολύ θαραλέο ακτιβιστή που συναντήσαμε στα πλαίσια της εκδήλωσης για το Ζαχάροφ. Τέλος πάντων θα συνεχιστούν οι επαφές με τις βραζιλιάνικες αρχές κάποια στιγμή κατά τα μέσα του έτους αλλά και με την ε, κοινωνία τους εκπροσώπους της δηλαδή. Επίσης μας είπατε για την Κούβα. Όχι, όχι, δεν συζητήσαμε μόνο για προστασία δεδομένων. Και αυτό είναι σημαντικό για το θέμα των γυναικών. Αλλά είπαμε ότι πρόκειται για θέματα που είναι αντικείμενο συνεργασίας. Οπότε στεκόμαστε σε αυτά ως αφετηρία και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων πιο αποτελεσματικά, στα πιο καυτά. Ε, βέβαια μιλήσαμε για τους πολιτικούς ε, κρατουμένους, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν αυτά και το Κοινοβούλιο γενικότερα για τις πολιτικές ελευθερίες για την ελευθερία στο Ιντερνετ, ελευθερία έκφρασης. Ήταν ε, μακροσκελής οι συζητήσεις μας. Κράτησαν πολύ τώρα για τη ΣΥΠΑ. Ναι, το μεταναστευτικό, η θανατική ποινή. Είπαμε ότι νιώθουμε απογοήτευση για τις ε, εκτελέσεις θανατική ποινή, μια που έχουμε την πρόσφατη απόφαση να εκτελείται θανατική ποινή για υποθέσεις ομοσπονδιακού χαρακτήρα και στην Ουάσιγκτον συνάντησα κάποιους φορείς ε, κοινωνικούς εκπροσώπους των πολιτών που ασχολούνται με την θανατική ποινή, τα είπαμε και επίσης συγκροτήθηκε κάποια επιτροπή στη χώρα για κάποια δικαιώματα που δεν μπορούν να απεμποληθούν και είπαμε ότι έχει αμερικανική απόχρωση το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί, είναι και θέμα συνταγματικό, αλλά και θέμα διεθνούς δικαίου. Και θα ήθελα να συναντήσω τον πρόεδρο της σχετικής ε, επιτροπής στην επόμενη αποστολή μου στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε όσον αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αποχώρηση. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με τη χώρα για αυτά τα ζητήματα και αυτό θα το προσέξω ιδιαίτερος. Για τη Σαουδική Αραβία που αναφέρθηκε από μια σειρά βουλευτών είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε. Κάτι, ο Φιλμπένιον, η Σαβέλη, η Άννα. Οπότε εκρεμεί η ιδέα του να τα συζητήσουμε με τη χώρα εδώ και ένα χρόνο ή περισσότερο και στη συνέχεια αυτού προσφέραμε κάποιες ευκαιρίες, κάποιες προτάσεις που κάναμε προς την χώρα. Ακόμα όμως δεν υπήρξε κάποια συνεννόηση. Σύμφωνα με τα όσο προτείναμε, είχαμε βέβαια προσκλήσει όπως και χθες μόλις για συζήτηση ανθρωπινών δικαιωμάτων και είπα ότι ναι, προτίθεμαι να πάω και να συμπροεδρεύσω κάποια εκδήλωση για διάλογο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει όμως να έχει νόημα αυτή η εκδήλωση. Ε, θα πρέπει να έχει επιφανειακό χαρακτήρα. Γιατί υπάρχουν ουσιαστικά θέματα. Η θανατική ποινή, οι εκτελέσεις που αυξήθηκαν πέρσι σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία και έχουμε και συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και υποθέσεις που τις ε, ανέφερα χθες τον Υπουργό ακτιβιστές που είναι φυλακισμένοι λόγω της δραστηριότητά τους και όλα αυτά τα συζητήσαμε. Θέλουμε να τα συζητήσουμε με τη χώρα, έχουμε και θέματα άλλα που αφορούν την Ευρώπη. Αναφέρθηκαν χτες, ε, εντάξει, αυτό θα πει διάλογος και χρειάζεται σοβαρή δέσμευση. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε γιατί η χώρα είναι σημαντική. Πάντως μέχρι τώρα δεν τα έχουμε βρει. και ανέφερες ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες και εσύ ναι θα πρέπει να αναβαθίσουμε τον ρόλο μας στα πολυμερή φόρα αφού αποχώρησαν από το Συμβούλιο εκείνη και θα πάω στην επόμενη συνεδρίαση στην ε, Γενέβη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου που θα γίνει τον Φεβρουάριο Ήδη προετοιμάζομαι. Πάντως θα πρέπει να συνεχιστούν οι, οι επαφές με τη χώρα. Επίσης αναφέρθηκε και η Ινδία. Τώρα δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, για να πάω στη χώρα, αλλά όπως αναφέρε οι βουλευτές που μίλησαν γι' αυτό, όταν πάω στο Πακιστάν θα είναι ευκαιρία να πάω και στην Ινδία και εγώ έτσι το προγραμματίζω. Βέβαια υπάρχει και το θέμα του Κασμίρ που αναφέρατε και θα συζητηθεί στα πλαίσια αυτών των επαφών τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κασμίρ που το ελέγχει η Ινδία αλλά και το Πακιστάν στο βαθμό που εμπλέκεται. Άρα θα γίνει συνεργασία για να δούμε τι θα κάνουμε με το πρόβλημα. Θα τα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε. Η Ισαβέλα, πρώτα-πρώτα, μπράβο. Συγχαρητήρια για την έκθεση για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαντική η δουλειά σου, αλλά μπράβο και στην Επιτροπή. Τώρα για αυτά που ρώτησες. Βιετνάμ και Βενεζουέλα. Και η πρόεδρος ανέφερε το Βιετνάμ. Για το Βιετνάμ. Υπάρχει ε, επαφή, υπάρχει διάλογος, θα τα ξαναπούμε μέσα Φεβρουαρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προβληματιζόμαστε για τη συμμετοχή μας πάντως στον διάλογο που ισχύει. Να δούμε σε τι επίπεδο από πλευρά Βιετνάμ θα γίνει αυτός ο διάλογος, οπότε πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία. Μπορεί να είναι υπουργικού επίπεδου. Οι ενδείξεις πάντως είναι μάλλον αρνητικές για αυτό το επίπεδο διαλόγου. Εγώ πάντως προτίθεμαι να κανονίσω μια αποστολική για διμερείς επαφές κάποια στιγμή φέτος. Έτσι θα συζητήσουμε κάποια θέματα που έχουν ε, προκύψει. Πάντως, στο πρόγραμμα του Βιετνάμ είναι και όσον αφορά τις επαφές στο ΑΣΕΑΝ εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σχετικό διάλογο. Επίσης, και εσείς κυρία Πρόεδρε, ρωτήσατε για το τι γίνεται με τις εμπορικές συμφωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι γενικόλογα θα μπορούσα να πω το εξή. Δεν συμμετέχω βέβαια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά θα μπορούσε να πει κανεί ότι καλύτερα να έχουμε εμπορικές συμφωνίες παρά να μην έχουμε. Έχουμε έτσι ε, κάποιο μέσο πίεσης για το μέτωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, βέβαια, όταν έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις της εμπορικές συμφωνίες, ακόμα πιο ισχυρό μέσο πίεσης έχουμε και μηχανισμούς. Πάντως, το να υπάρχουν οι συμφωνίες και σχετική δραστηριότητα μας ισχυροποιεί την θέση στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βενεζουέλα. παρακολουθώ τις εξελίξεις. Έγινε και η σχετική διάσκεψη τον Σεπτέμβριο και παρακολουθώ το τι κάνει η Διεθνής Ομάδα Επαφής, ο ειδικό απεσταλμένος. Ξέρω τις σχετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις που έχουν γίνει πρόσφατα. Εννοείται ότι είναι πολύ προβληματική κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας προβληματίζει και λέω να πάω τον Φεβρουάριο στην Κολομβία. Και έχουμε πολλούς ε, μετανάστες και στην Κολομβία και σε άλλες γειτνιάζουσες χώρες, οπότε και αυτό είναι ένα από τα ζήτηματα που θα μας απασχολήσουν. Χάουταλα μας είπες για τις ε, κυρώσεις. Πώς έχει κατάσταση. Ευτυχώς. Δεν χαράζω εγώ την πολιτική, αλλά φροντίζω για την εφαρμογή, άπαξ και τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα αποφασίσουν σχετικά. Εννοείται ότι και εγώ βάζω το χεράκι μου με το που εξελίσσονται οι πολιτικές ε, έχω τις παρατηρήσεις μου και κλήθηκα στο Συμβουλίο Εξωτερικό όταν συζητήθηκαν οι κυρώσεις υπήρχε ευρεία συνένεση θεωρήθηκαν σκόπιμες οι κυρώσεις υπήρχε και ένα non-paper Αυτό το non τώρα συζητείται από τα κράτη-μέλη. Και να δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Ε, εννοείται ότι είναι άλλο ένα όπλο, άλλο ένα μέσο πίεσης οι κυρώσεις ε, σε σχέση με το θεματολόγιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακολουθώ τις εξελίξεις από κοντά. Άλλο. κυρία Χάουταλα επίσης αναφέρει το θέμα τη σχέση ε, επιχειρήσεων και η επιχειρηματικότητα τέλο πάντων και δικαιωμάτων σε σχέση με τις επαφές ε, με την Αφρικανική Ένωση. Ναι, ήταν ένα τομέα που προχωρήσαμε στις συζητήσει. είχαμε κάποιες εκδηλώσεις όπου θα συμμετέχουν και οι δύο πλευρές. Υπήρξαν και κάποιες αποκλήσεις απόψε με κάποιες αφρικανικές ε, χώρες. Είχαμε αυτό το δεσμευτικό μέσο πολιτικής. Το είδαμε στην Γενέβη. Τι γίνεται με, τις, ε, με την διεθνή συνεργασία. Και το θέμα αυτό για το δεσμευτικό μέσο νομίζω ότι προσφέρεται σε αυτό το μέτωπο έδαφος ε, πρόοδου. Υπάρχει προοπτική πρόοδου και είπαμε ότι έχουμε 26 χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτή την υπόθεση 13 ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τις βασικές αρχές το θέμα της δέουσας επιμέλειας που αναφέρατε και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης ε, και πρέπει να προχωρήσουμε και προς τα εκεί. Πάντως θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσω περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί νομίζω ότι σε κάποιες από τις εκδηλώσει που πήγα συζητήθηκαν όλο ένα και περισσότερο υπάρχει προβληματισμός από πλευρά εταιριών, επιχειρήσεων. Σχετικά με αυτό, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα τι ζητούν οι πελάτες των επιχειρήσεων, το ξέρουν οι επιχειρήσεις. Τι ζητούν οι καταναλωτές που όλα και περισσότερη ευαισθησία έχουν για την υπόθεση των δικαιωμάτων. Οπότε από πλευρά του πολιτικού κόσμου, των θεσμικών οργάνων, ε, των διπλωματικών φορέων, το ξέρουμε. Α, και θα πρέπει βέβαια να δούμε τι γίνεται στις επαφές μας με τις επιχειρήσεις. Παλαιστίνη, ναι, ξέρουμε. Εκεί τι καταπτώσεις δικαιωμάτων γίνονται. Πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα και στη Γάζα. Έχουμε και την εκτόξευση των πυράβλων από Γάζα προς Ισραήλ που και αυτό προβληματίζει. Θέλω να κάνω μια αποστολή σε Παλαιστίνη και Γάζα. Και έχω μιλήσει με τους ομολόγους μου, τους, με τους συναδέλφους που μας αντιπροσωπεύουν εκεί σε αυτά τα μέτωπα, με την Σουζάνα που είναι εκεί και ίσως από κοινού ε, κάνουμε κάποια κίνηση φέτος. Ε, μισό λεφτάκι τώρα. Να ρίξω μια ματιά στις σημειώσεις. Α, η Νταϊάν. Τέθηκε το θέμα... Να, έφυγε η Νταϊάννα. Θα απαντήσω όμως. Τέθηκε το θέμα της συνέπειας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού. Θέλω να είμαι σαφής εδώ. Η εντολή μου, τα καθήκοντα που έχω αναλάβει, έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, εκτό Ένωση. Είμαι ο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να επεξηγήσουμε εδώ ότι μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εξωτερική δράση της Ένωσης. Εντάσσεται στα πλαίσια εξωτερικής μας πολιτικής δηλαδή αυτό που κάνω. Βεβαίως πρέπει να έχω συνείδηση του τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δουλειά μου. Πρέπει να είμαστε συνεπείς το τι κάνουμε εντός των τυχών και τι κάνουμε εκτός. Διότι όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, υπάρχουν χώρες με τις οποίες ε, συζητούμε για ανθρωπινά δικαιώματα και οι οποίες άμεσα μας λένε πολύ γρήγορα και σωστά ότι ξέρετε και εσείς έχετε προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τάδε ή στο δίνα κράτος μέλος. Είναι λογικό να το κάνουν αυτό είναι κάτι το οποίο καλωσορίζω μάλιστα σε συζητήσει με τρίτε χώρες, διότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει ειλικρινή διάλογο και είναι και ρόλος μου ε, να το αναφέρω αυτό στη συνέχεια εδώ, σε εσωτερικό επίπεδο και ότι πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα. Είχα πάει στη Βιέννη να συζητήσω με την η Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων, όπως σας είπα, πολύ σημαντική συνάντηση, διότι εκεί έχουμε μια εικόνα του ποια είναι η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει έρευνα, υπάρχει αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την απόδοση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τη Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων. Έχουν, υπάρχει δηλαδή μεγάλος όγκος έρευνας. Παραδείγματο χάρη για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση ή την θέση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που είναι ζητήματα κράτους δικαίου ε, μεταξύ άλλων. Πρόθεσή μου είναι λοιπόν να βασιστώ σε αυτά που μας λέει η Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων της Βιέννης. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα συμμετείχαν αξιωματούχοι από αυτήν την υπηρεσία ε, στον διάλογο που είχαμε Ε, είναι ένα γενικό ζήτημα αυτό για τα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκουν σε κάποια χώρα ή σε κάποια ήπειρο. Είναι αφορούν το σύνολο της υφηλίου. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό και να το θυμόμαστε ε, πάντα. Ε, βεβαίως κάποιες χώρες θα πάνε καλύτερα από άλλες. Αλλά καμία χώρα δεν έχει λευκό ποινικό μητρό ε, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στι τρίτε χώρε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εμεί δίνουμε μία εικόνα ότι ερχόμαστε και δίνουμε μαθήματα. Ερχόμαστε με τι ευρωπαϊκέ μα αξίε και αυτό και εκεί συχνά υπάρχει μια πρόσληψη ε, της δράσης μας αυτής ως μια νεοαπικιακή ε, προσέγγιση. Η δική μου προσέγγιση λοιπόν εδώ είναι πάντα να θυμάμαι από πού ερχόμαστε, έτσι. Να μην ξεχνάμε την ιστορία αυτής της Υπήρου. Και πώς ε, στα μέσα του 20ου αιώνα η συνεισφορά μας στην δομή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, έρχεται μετά από μια ιστορία Πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί. Βεβαίω, ορισμένε φορέ υπάρχει μια διασύνδεση. Ορισμένε φορέ ε, δεν δίνουμε επαρκή σημασία, παραδείγματο χάρη, στα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα. Επικεντρωνόμαστε σε μεγάλο βαθμό ε, σε, στα πολιτικά δικαιώματα και σωστά, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν και σε άλλους τομείς. Λοιπόν, τι μου έχει μείνει εδώ. Δεν ξέρω αν μου λείπει κάτι. Ναι, τέθηκε ένα ερώτημα ενδεχομένω για τις μελλοντικέ μας συνεδριάσεις είναι δύσκολο να δημοσιεύουμε το πρόγραμμα διότι ε, ως και την τελευταία στιγμή αλλάζουν αυτά. Αλλά το είπατε και την προηγούμενη φορά του Σεπτέμβριο ότι πρέπει να θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητε μου. Έκτοτε περιοδικά δημοσιεύω ε, ένα δελτίο με μια περίληψη όχι όλων όσων κάνω αλλά τα, των πλέον σημαντικών. Ε, θα μπορούσε αυτό ε, να βοηθήσει στο μέλλον. Ε, ενδεχομένως και η Επιτροπή να μας πει, να μου πει αν υπάρχουν κάποιες θεματικές με τις οποίες θέλετε να ασχοληθώ ε, θα ήταν καλύτερο αυτό από το να έχετε με πλήρη αναφορά όλων αυτών που κάνω. Συγγνώμη αν ξέχασα να απαντήσω σε κάποιον, ευχαριστώ να επανέλθω. Ευχαριστώ Ήμων. Ναι, είναι ενδιαφέρον να αρχίσαμε έτσι τη χρονιά με μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας ε, αλλά αυτή η ιδέα να σας καλούμε σε αυτή την επιτροπή ε, για να συζητήσουμε συγκεκριμένες θεματικές είτε γεωγραφικές ε, είτε για συγκεκριμένα ζητήματα είναι μια καλή ιδέα θα το λάβουμε υπόψη μας λοιπόν στα πλαίσια συνδυασία των συντονιστών όταν θα σας καλέσουμε την επόμενη φορά ποιες θα μπορούσαν να είναι θεματικές που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε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 On Σας ευχαριστώ όλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο της διάταξης. Το επόμενο σημείο για την Μιαμάρ. Θα ήθελα παρακαλώ να καθίσετε Χαίρομαι που συμπροεδρεύω το σημείο αυτού με τη συνάδελφο τη Μάριαν Βίντ, αντιπρόεδρο τη αντιπροσωπεία για τι σχέσει με τι ε, χώρε τη Ασίας, της Νοτιοανατολικής Ασίας και με την Ένωση των Εθνών τη Νοτιοανατολικής Ασία ε, πάντα συμμετέχουν οι των αντιπροσωπιών έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέπεια σε ό,τι φορά το έργο μας για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για του Ροχίνγκια. Ροχίνγκα. Από το 2018 πήγε μια αντιπροσωπεία μα στη Μιαμάρ. Πρόσφατα υπήρξε μια επίγουσα, ένα επίγον ψήφισμα του Κοινοβουλίου ε, για την κατάσταση στη Μιανμάρ, ιδιαίτερα την κατάσταση των Ροχίνγκα. Ε, έρχεται με στη συνέχεια δύο ακόμα ψηφισμάτων από το 2015. Μια από τι βασικέ ανησυχίε μα είναι η αντιμετώπιση τη ατιμορρησία και τη ευθύνη για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ατιμορρησία πουθενά. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεστροποιηθεί στο ζήτημα αυτό. Όπω γνωρίζετε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δύο μηχανισμού που επιτρέπει έρευνα για τι ενδεχόμενε παραβιάσει των δικαιωμάτων στη Μιαμάρη. Πρώτο, πρώτο ήταν η ανεξάρτητη διεθνή αποστολή για να δούμε ποια είναι τα γεγονότα, τα, τα συμβάντα, ε, σε ποιε προποθέσει έλαβαν χώρα ε, παραβιάσει των δικαιωμάτων από το στρατό και βεβαίω να συλλέξει πολιτικά στοιχεία. Παρουσιάστηκαν συμπεράσματα και συστάσει στην τελική τη έκθεση το Σεπτέμβριο του 2019 στο Συμβούλιο των Δικαιωμάτων και ολοκλήρωσε εκτέκτοτε την ε, εντολή τη. Ο δεύτερο μηχανισμό είναι ο, μηχανισ... ο ανεξάρτητο μηχανισμό έρευνα των ΗΕ για τη Μιαμάρ που δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018, που μόλι έχει ξεκινήσει τι δραστηριότητέ του μια και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2019. Θα προετοιμάσει φακέλου για να διευκολύνει και να επιταχύνει ποινικέ διαδικασίε ανεξάρτητε και ε, δίκαιε. Και βεβαίω θα βασιστεί στα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανεξάρτητη έρευνα. Ε, η διεθνής, ε, το Διεθνές Δικαστήριο έχει ε, ξεκινήσει την ε, εξέταση τη υπόθεση που έχει προσφύγει η Γκάμπια κατά της Μιαμάρ, ότι η Μιαμάρ δηλαδή δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της ε, σύμφωνα με τη σύμβαση του 1948 για την ε, πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκλημάτων γενοκτονία. Ε, έκτοτε υπάρχει η προσπάθεια να υπερασπιστεί το δικαίωμα τη χώρα της Πρωθυπουργό της Μιαμάρ. Ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, θα εξεταστεί το ζήτημα και θα εξεταστούν βεβαίως και οι ατομικές ε, ποινικέ ευθύνες. Τον Νοέμβριο του 2018 ε, ο εισαγγελέα του δικαστηρίου ξεκίνησε μία έρευνα στα σύνορα μεταξύ Μιαμάρ και Μπαγκλαντές. Η κατάσταση λοιπόν είναι εν εξελίξη από το 2015 μας απασχολεί εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε προλέσει την ανταλλαγή απόψεων με τον Νίκολας Κούμιαν που είναι υπεύθυνο για τον ανεξάρτητο μηχανισμό έρευνας των ΗΠΑ για τη Μιαμάρ είναι εδώ μέσω web streaming μαζί μας και βεβαίω είναι εδώ και μαζί μας η Γιασμίν Ουλά τη ελεύθερη ε, Συμμαχία των Ροχίνγκα θα ξεκινήσουμε από τον προσκεκλημένο μας εξ αποστάσεως τον Νικόλας ε, Κούμιαν και στη συνέχεια δώσουμε το λόγο στην Γιασμίν για να δώσω συνέχεια στην συζήτηση. Έχετε το λόγο, εκτός εάν θέλει να προσθέσει κάτι η, η συνάδελφος εδώ, η Μάριαν, στην εισαγωγή της. Ναι, βεβαίω αναμένω με την υπομονησία να ακούσω τις ομιλίες αυτές. Ε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχουμε φτάσει το 2020 ε, και ακόμα ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Συμμετέχω και στην ομάδα των Ευρωβουλευτών ε, που ε, το Μάιο θα επισκεφτεί την περιοχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκεί με όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ Μάριαν. Νίκολας έχετε το λόγο. Ε, Έχει... Ακούτε, έχετε μετάφραση, πολύ ωραία. Εντάξει, στα αγγλικά και όλοι καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ. Ονομάζομαι Νίκολα Κουντζιάν και είμαι επικεφαλή του ανεξάρτητου μηχανισμού έρευνα ε, για την Μιανμάρ. Ε, και ευχαριστώ τα μέλη της Υποεπιτροπής για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για το όσα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν σημαντικά τον μηχανισμό και οφείλουμε πολλά σε εσά. Ο μηχανισμός να γνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τακτές επαφές και θα συνεχίσουμε να στηριζόμαστε και να υπολογίζουμε σε αυτήν την βοήθεια. Για να δούμε τώρα λίγο το ιστορικό πλαίσιο τον Σεπτέμβριο του 18, όπως αναφέρατε. Είχαμε αυτή την ερευνητική των πραγμάτων αποστολή στη Μιανουμάρ και αναφέρθηκε ότι υπήρχαν ε, ε, στοιχεία βάσιμα ούτως ώστε να τεκμηριώνονται κάποια σοβαρά εγκλήματα τα οποία είχαν ε, διαπραχθεί και να σταματήσει η ατιμορρησία. Μετά είχαμε το ψήφισμα 39 ε, κάθετος 2 και ε, έτσι ο μηχανισμός μας συγκροτήθηκε ούτως ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε, να ε, προστατεύσουμε τα στοιχεία που υπήρχαν για τα πιο σοβαρά από αυτά τα εγκλήματα και παραβιάσεις του εθνούς δικαίου. Και η εντολή μας ήταν και παραθέτω να προτιμάσουμε τον φάκελο ώστε να διευκολύνουμε και να διεκπεριώσουμε τη σχετική ανεξάρτητη ποινική διαδικασία σύμφωνα με τα πρώτα του διεθνούς δικαίου σε επίπεδο διεθνών περιφερειακών ή διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων που θα έχουν την δικαιοδοσία σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας από κοινού υποστήριξαν αυτήν την συγκρότηση του διοδυτικού οργάνου.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 Just, just one minute, Μισό λεπτό, Νίκολας. Λέει η πρόεδρος. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο. Υπάρχουν τόσες παρεμβολές που δεν ακούγεσαι καλά. Μήπως μπορεί κάποιος τεχνικός να το ρυθμίσει. <laughs>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 as we move forward into implementing, further implementing our very difficult mandate. Thank you again for this opportunity to brief the subcommittee, and I welcome your questions. Thank you. Thank you, Nicola. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκολας, για την παρουσίαση αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και φαντάζομαι θα τεθούν και αρκετά ερωτήματα. Δίνω όμως πρώτα το λόγο στη Γιασμίν Ουλά και μετά θα δώσω το λόγο τους ε, ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Η Γιασμίν, λοιπόν, έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. Honorable members of... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ε, αγαπητοί ε, φίλοι, Χαίρομαι που μου δώσατε τη δυνατότητα να έρθω σήμερα εδώ, αλλά η παρουσία μου εδώ ε, με επιβαρύνει και εμένα ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ε, βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο, ε, αλλά η πλειοψηφία του λαού μου συνεχίζει να ζει με φόβο και να υποφέρει. Ο φόβος είναι μια εμπειρία πάρα πολύ συνηθισμένη που προσδιορίζει το ποιοι είμαστε ως Ροχίνγκια. Ανεξάρτητα από το φύλλο μας, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, ο φόβος είναι στενά ε, συνειφασμένος με την ύπαρξή μας. Μετά από δεκαετίες διώξεων, ο πόνος που μας έχει επιβληθεί από τη στρατιωτική εξουσία στην ε, Μιανμάρ ε, μας κάνει να νιώθουμε αβοήθητοι και παγιδευμένοι. Σχεδόν ε, όλοι οι Ροχίνγκια έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους νιώσει αυτό το συνέστημα. Εγώ το ένιωσα όταν ήμουν πρόσφυγας στην Ταϊλάνδη χωρίς καθόλου προστασία και θυμάμαι προσευχόμουν κάθε μέρα να γυρίσουν ασφαλείς πίσω οι γονείς μου που προσπαθούσαν να βγάλουν τα προστοζήν πουλώντας ε, στο, στο δρόμο ε, κάτι για να συνεισφέρουν το φαγητό της οικογένειας. Εκείνη την εποχή ε, προσευχόμουν τη στιγμή που μπαίναμε Έμπαινα σε ένα κελί στο ε, τμήμα ε, μεταναστών ε, της Ταϊλάνδης γιατί μας είχαν σε ένα κέντρο κράτησης επειδή δεν ήμασταν νόμιμα στην Ταϊλάνδη. Προσευχόμουν να μην μας εκτοπίσουν στη Μιανμάρ και δεν είχα προσευχηθεί ποτέ τόσο πολύ στη ζωή μου όσο τότε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξεφύγει κανείς από αυτή την κατάσταση όταν είναι ροχίνγκια. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια στιγμή που να μας μεταχειρίζονται με σεβασμό, σαν να είμαστε πραγματικά ανθρώπινα όντα. Φόβο ένιωθαν τα αδέρφια μου που ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες στο Μπαγκλαντές, σε στρατόπεδα και που ζουν ακόμη οι ε, συμπολίτε μου σε στρατόπεδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ο φόβος ισχύει και για αυτούς που ζουν ε, σε συνθήκες περιοριστικές στη Μιανμάρ. Ισχύει για όλους αυτούς ε, που ζουν σε κάποια από τις χώρες ΑΣΕΑΝ και φοβούνται ότι θα συλληφθούν κάποια στιγμή ακριβώς επειδή είναι ροχίνγκια. Ε, γιατί ενώ παλιότερα συνεισφέραμε στην οικονομία της Μιανμάρ, καταλήξαμε να είμαστε πρόσφυγες, παράνομοι, boat people. Μας ανάγκασαν να δεχτούμε κάτι που είναι πολύ πολύ λιγότερο από αυτό που αξίζει πραγματικά ένα ανθρώπινο όν. Και αυτό είναι κάτι που μας καταστρέφει την αίσθηση ε, του ανθρώπου το θέμα της ηθαγένειας των Ροχίνγκια, η, η αρχή του αγώνα μας που έχει κρατήσει εδώ και δεκαετίες, ε, μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ απλό, ιδίως ε, στην κυβέρνηση της Μιανμάρ, τη μη στατιωτική κυβέρνηση, που ε, επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται μια επαλήθευση της ηθαγένειας του λαού μου. Ήδη και στο Διεθνές δικαστήριο τον περασμένο μήνα επανέλαβε ε, αυτή την ε, αφήγηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας ε, η ηθαγένεια, για μας στην περιφέρεια του Ράκιν που είμαστε θύματα καταπίεσης και δράσεων εκαθάρισης από τους στρατιωτικούς και όλα αυτά γίνονται σε επιδίωξη έργων οικονομικής ανάπτυξης και κονδυλίων από τις διάφορες γειτονικές χώρες όπως ε, η Ιαπωνία, η Κίνα και άλλες. Όσο περισσότερο ανοίγεται η χώρα σε επιχειρηματικές κινήσεις, τόσο περισσότερο υποφέρουν οι Ροχίνγκια και άλλες εθνοτικές ε, μειονότητες. Οι επενδύσεις και οι επιχειρηματικές συνεργασίες έχουν βοηθήσει τις διάφορες κυβερνήσεις και τις στρατιωτικές αρχές στη Μιανμάρ να παραμείνουν στην εξουσία παρά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρά της γενοκτονίας. Πριν από λίγες μέρες, το γραφείο της Προεδρίας της Μιανμάρ εξέδωσε μια έκθεση της αποκαλούμενης ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας, επαναλαμβάνοντας αυτά που έλεγαν οι στρατιωτικοί και οι δικτάτορες στη Μιανμάρ. Και αντί να κατηγορεί την αστυνομία και τις δυνάμεις εξουσίας, προσπαθούν να εξοραίσουν την κατάσταση μιλώντας ε, για βία μεταξύ κοινοτήτων για τους Ροχίνγκια. Επίσης, ε, ε, λέει ότι οι μαζικοί βιασμοί ήταν απλώς αβάσιμοι ισχυρισμοί χωρίς να έχει πάρει συνέντευξη από κανένα από τα θύματα που ζουν σε στρατόπεδα. Και ειλικρινά όταν είδα αυτό το τμήμα της ε, έκθεσης πραγματικά πόνεσα, γιατί αυτό δείχνει τις πατριαρχικές απόψεις που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά και διονίζονται από την κυβέρνηση, ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο. Και για μας δείχνει και για μας και σε άλλες εθνοτικές μειονότητες, δείχνει ότι η ατιμορρησία είναι πιο σημαντική για την κυβέρνηση της Μιανμάρ από το να υπερασπίζονται τις γυναίκες και τα κορίτσια που βιάστηκαν στη χώρα μας. Αναφέρθηκαν ε, ως ε, ένστικτο προστασίας σε περιπτώσεις βίας μεταξύ κοινοτήτων αυτά τα οποία έγιναν και οι τεράστιοι αριθμοί ροχίνγκια που έφυγαν από τη χώρα ως πρόσφυγες ε, υποτίθεται ότι δρούσαν με βάση αυτό το ένστικτο προστασίας. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι οι μητέρες δεν θα έβαζαν ποτέ τα παιδιά τους στον κίνδυνο να πνιγούν περνώντας ένα ποτάμι αν υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού τους. Η αποκαλούμενη Επιτροπή Έρευνας κατέληξε στο ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη συμπεριφοράς που θα μπορούσε κανείς να πει ε, ότι ε, διαπράχθη με πρόθεση γενοκτονίας. Ε, λέγουν ότι οι αντιδράσεις των ε, δυνάμεων ασφαλείας πηγάζουν από το φόβο τους, από βαθιά ριζωμένες διαφορές μεταξύ των ε, κοινοτήτων και οι στρατιωτικές δυνάμεις εξεπλάγησαν και αντέδρασαν έτσι. Και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ακούσει τέτοιες ιστορίες πολλές φορές. Υπερασπίζονται τα βία εγκλήματα κατά του λαού μου και έχουμε πολλές μαρτυρίες που μπορούν να το διαψεύσουν αυτό. Η Ρακιούμα που έφυγε ως πρόσφυγα στο Μπαγκλαντές ε, ε, ε, το 2017 διηγείται την ιστορία, της, την ιστορία του γιού της, ένα μωρό που της το πήραν από τα χέρια και το πέταξαν στη φωτιά. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες ιστορίες που τα παιδιά τα πήραν από τα χέρια των γονιών τους και τα σκότωσαν δεν εξεπλάγησαν οι στρατιώτες τη στιγμή εκείνη, έδρασαν προγραμματισμένα και με βιαιότητα, προσπαθώντας να αποσταθεροποιήσουν οποιαδήποτε αίσθηση κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τον τοξικό χαρακτήρα των εκτελεστικών δυνάμεων. Επιβεβαιώνονται οι υποψίες ότι οι τωρινοί θεσμοί και οι θύνοντες δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν και δεν προσπαθούν να κάνουν τη χώρα πιο δημοκρατική, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και κάτι που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι μεγαλύτερη υποστήριξη. Θα ήθελα να επικεντρωθείτε στη δράση των ακτιβιστών επιτόπου, των νέων της Μιανμάρ, που παλεύουν εναντίον όλων αυτών των αφηγήσεων μίσους που πηγάζουν από την προπαγάνδα των στρατιωτικών. Αυτοί οι άνθρωποι επιτόπου, αυτοί οι νέοι, είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή και αυτοί χρειάζονται πάρα πολύ τη βοήθειά σας και την προστασία από το καθεστώς καταπίεσης. Δεδομένου ότι οι θύνοντες δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν, πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να επανεξετάσει τις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες ή το EBA, το όλο εκτός από όπλα, εφόσον ο κανονισμός των γενικευμένων προτιμήσεων ορίζει ότι εμπορικές προτιμησιακές σχέσεις μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού η Μιανμάρ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, παραβιάζει αυτές τις αρχές επανειλημμένα και ίσως τώρα πρέπει οι στρατιωτικοί να καταλάβουν ότι δεν θα επωφεληθούν, δεν θα ξαναπάρουν ούτε ευρώ από τέτοιες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, όσο συνεχίσουν να διώκουν αθώους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μιανμάρ. Οι θεσμοί στη Μιανμάρ έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την πραγματικότητα για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τη θέση της Μιανμάρ παγκοσμίω, προσπαθώντας να δείξουν ότι όλο πάνε καλά στη χώρα. Και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν εσωτερικά. Είμαι εδώ σήμερα για να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα του να εξετάσουμε τις παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστηματικά. Παράλληλα, είμαι εδώ για να κάνω έκκληση στη συνείδησή σας ε, ως ανθρώπινο όν. Ο λαός μου δεν ζητάει ένα χωριστό κράτος, δεν ζητάμε μια πολυτελή ζωή. Δεν ζητάμε τίποτα το ακατόρθωτο δεν ζητάμε τίποτα που να μην μπορείτε να το επιτύχετε. Συνεχίζουμε να υψώνουμε τη φωνή μας για να μπορέσουμε να ακουστούμε, για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από αυτό το αίσθημα του ότι είμαστε αβοήθητοι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Είναι υπερβολικό αυτό το αίτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κατάλληλος φορέας γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ζήσει τη γενοκτονία και τις μαζικές βιαιότητε. Γι' αυτό έχουμε και την Σύμβαση για τη Γενοκτονία. Και άλλοι μηχανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκίνησαν από εδώ. Και θα πρέπει όλοι εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσετε ε, αυτά που έχετε στη διάθεσή σας ως εμπειρία και να ζητήσετε ε, κάποια καλύτερη τύχη για τα θύματα των εγκλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί την προσφυγική κρίση και θα ήθελα να συζητήσω ζητήσω μεγαλύτερη ενίσχυση και μεγαλύτερη υποστήριξη προς τη χώρα που μας υποδέχεται, τον Μπαγκλαντές. Δεν θα πρέπει τον Μπαγκλαντές να νιώθει εγκαταλειμμένο μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τέλος, το Διεθνές Δικαστήριο θα διαβάσει την απόφασή του αύριο. Ανεξάρτητα όμως από την απόφασή του, εγώ και η κοινότητά μου ελπίζουμε πραγματικά ότι θα συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε. Ότι θα συνεχίσετε να βρίσκεστε στο πλευρό μας και να προωθείτε μέτρα λογοδοσίας και δικαιοσύνης που τα χρειάζεται τόσο πολύ η Μιανμάρ. Η χώρα μου, στην οποία τυραννικές κυβερνήσεις και στρατιωτικές διοικήσεις κυβερνούν το λαό. Θέλουμε να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας από το λαό και για το λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you. Thank you very Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους ευρωβουλευτές. Ξέρετε πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση Έχουμε ένα τέταρτο μόλις. Είναι λίγο ο χρόνος. Οπότε σα παρακαλώ να είστε σύντομοι ε, στις παρεμβάσεις και να περιοριστείτε ουσιαστικά σε ερωτήσεις. Η Ιζαμπέλ δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς μετά από αυτά που μόλις ακούστηκαν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Είπατε αυτά που έπρεπε να υποθούν ε, και πρέπει να είστε βέβαιοι ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Κύριε Κόμιαν, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς ε, τη δυνατότητα με βάση ε, την παρούσα κατάσταση ε, να βελτιωθούν τα πράγματα στη Μιαμάρα. Αυτή η έρευνα έχει κάποιο αντίκτυπο ή όχι. και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να προχωρήσει αυτή η έρευνα. Ήθελα επίσης να ρωτήσω η κοινή γνώμη της Μιανμάρ πώς αντιδράει σε αυτά που συμβαίνουν στους Ροχίνγκα. Εμείς ως Ευρωπαίοι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσω στα γαλλικά, συγγνώμη είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από τις εξελίξεις στη Μιανμάρ. Δεν το περιμέναμε αυτό πριν από μερικά χρόνια. Ορισμένε φορέ έχω την εντύπωση ότι ε, έχουμε και εμεί ευθύνη. Ε, σταματάω γιατί πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Πραγματικά σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη μαρτυρία σα και για το έργο που κάνετε εσείς με τον μηχανισμό αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ, Ιζα, Ιζαμπέλ τώρα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Το πρώτο μου ερώτημα είναι για τον ε, συνομιλητή μας εδώ στη Γενέβη, ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι κεντρικές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε για να μπορέσετε να συλλέξετε αποδεικτικά στοιχεία για γενοκτονία. Επίσης, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε για να, για να εγγυηθείτε την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Και ένα ερώτημα για τη Γιασμίν. Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε επί τόπου για να έχετε πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είναι προφανές ότι εκεί όπου ζείτε δεν έχετε αυτή την πρόσβαση. Έχετε την εντύπωση όμως ότι οι διεθνείς αρχές έκαναν όσα έπρεπε για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην δικαιοσύνη και για να μπορέσετε να αποζημιωθείτε για όλες αυτές τις ιδεχτείς πράξεις. Ναι, συμμετέχω εδώ και δύο χρόνια στην προσπάθεια αυτή υπό άλλη ιδιότητα. Βλέπετε ότι εδώ, από ό,τι φαίνεται, εδώ εξετάζονται τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην περίοδο έως την Μεγάλη Έξοδο ε, πιο πρόσφατα όμως εμείς θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να εγγυηθούμε μια ασφαλή επιστροφή δεν έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προοπτική ασφαλούς επιστροφής παρότι τον, τον Παγκλαντές και Μιαμάρ διμερός προσπαθούν να βρούνε κάποιον τρόπο για να συμβεί αυτό είστε σε θέση να αξιολογήσετε ε, το κατά πόσο πληρώνται προϋποθέσεις για ασφαλή επιστροφή. Κατά τη γνώμη μου, εάν δεν υπάρχει επιστροφή της γης, ε, εάν δεν ε, υπάρξει ανοικοδόμηση των κατοικιών, ε, είναι δύσκολο. Υπάρχει κάποια πολιτική διαδικασία που να μπορεί να ακολουθηθεί και για το θεμελιώδη ζήτημα τη ηθαγένεια. Στη δική μας, στο δικό μα ψήφισμα το 2017 θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το θεμελιώδε, Ότι δεν έχουν δηλαδή ηθαγένεια σε μια Μάρη Ροχίνγκια, ότι του την αρνούνται. Ότι αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, διότι αυτό σχετίζεται και με την κατοχή γη και οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε λοιπόν να πάμε πέρα από τα εγκλήματα του παρελθόντος, διότι υπάρχει και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ε, των κέντρο προσφύγων στο Κόξις Μπιζάρ ε, οι αρχές του Μπαγκλαντές ε, θα δυσκολέψουν τη ζωή των ανθρώπων των προσφύγων εκεί ε, γι' αυτό είπατε ενδεχομένω και εσείς για την βοήθεια που να στην Μπαγκλαντές γιατί το Μπαγκλαντές προσπαθεί τώρα να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους ε, για να εκδιώξει τους ανθρώπους αυτούς και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ε, κόβεται το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα, δεν υπάρχει εκπαίδευση, παιδεία εκεί, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ε, βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα και την ID είναι ευχαριστώ μιλώ στο όνομα των πράσινων η Heidi. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας ε, κύριε Κούμιαν. Ε, κάνετε μια δουλειά η οποία είναι πολύ σημαντική και αξιόπιστη. Ευχαριστώ και η κυρία Ούλα για την ε, πολύ θαραλέα της δήλωση εδώ. Μας υπενθύμησε ε, βεβαίως και την κληρονομιά την ευρωπαϊκή σε επίπεδο γενοκτονίας. Δεν θα υπήρχε ενδεχομένως ε, σύμβαση για τις γενοκτονίες αν δεν είχαν λάβει χώρα αυτά που έλαβαν χώρα εδώ ε, και αν δεν είχαν αντιμετωπιστεί από τη διεθνή δικαιοσύνη. Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να εγγυηθεί την πρόσβαση ε, στην έρευνα της έρευνας, μάλλον όπου χρειαστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι από κοινού. Επίσης, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα περιορισμού σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική πρόσβαση στην περιοχή και πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, διότι από ανθρωπιστικής πλευράς τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα εκεί. Επίσης, ε, όντως, οι προτιμουσιακές εμπορικές συμφωνίες εξετάζονται εκ νέου αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς κυρία Ούλα. Ε, νομίζω ότι ο εισηγητής ε, για το διεθνές εμπόριο έχει αυτή τη στιγμή αποκλείσει το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Το παρακολουθούμε λοιπόν. Η Κομισιόν προφανώ και θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, διαδικασία αυτή. Τέλος, ε, το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει βεβαίω και του Ροχίνγκα, αλλά τότε δεν αναφέρθηκε η ευθύνη των ευρωπαϊκών εταιριών που βρίσκονται εκεί που είναι σε επαφή, κάνουν business με τις κρατικές αρχές, με το στρατό, χωρίς να μην, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει και αυτό το κομμάτι ε, να το φωτίσουμε κάπως, να το τονίσουμε, να το αναδείξουμε αυτές οι εταιρείε οι οποίες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Ναι, ευχαριστώ. Ε, είναι πολύ σημαντικό ότι το θέμα αυτό ε, έχει φτάσει στα δικαστήρια. Ε, είναι φοβερά αυτό που μας επιβεβαίωσε η κυρία Ούλα. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι η ζωή σας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει αυτή η βούληση επιστροφής στη Μιαμάρ από τον Μπαγκλαντές μετά από απόφαση του δικαστηρίου ή φοβάται ο κόσμος να επιστρέψει. Ευχαριστώ. Η πρώτα η Γιασμίν και μετά θα δώσω λόγο στον Νίκολας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το ερώτημά σας. Είναι περίπλοκο. Είναι περίπλοκη υπόθεση αυτή. Όταν μιλάμε για τραύματα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τραύματα τα οποία μας αφορούν σχεδόν όλους. Όλοι νιώθουμε ότι υπάρχει αυτός ο φόβος της επιστροφής σχεδόν όλοι όμως, όλοι μας θέλουμε να επιστρέψουμε. Και αυτό δείχνει το πόσο δεμένοι είμαστε με τα σπίτια μας. Βεβαίως άκουσα μαρτυρίες ε, γυναικών ε, που είδαν όλη την οικογένεια να δολοφονείται μπροστά στα μάτια τους, ε, τα παιδιά τους οι σύζυγοί τους, αυτές οι γυναίκες λένε θέλω να γυρίσω, θέλω να γυρίσω για να δω ακόμα και το τόπο εκείνο που σκοτώθηκαν, για να τους θυμηθώ. Από εκείνη τη μέρα και μετά είναι σαν να μην ζουν πια. Θέλω να επιστρέψουν λοιπόν εκεί όπου πέθαναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι τους. Είναι το τελευταίο πράγμα στο οποίο μπορούν να αγκιστρωθούν. Όσο και να θέλουμε βεβαίως να επιστρέψουμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο φύγαμε. Είχαμε πολλές εξόδους, μαζικές εξόδους τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Εγώ είχα φύγει το 1992 και είχαμε πολλές άλλες τέτοιες μετακινήσεις για να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, να υπάρξει κάποιος μηχανισμός δικαιοσύνης, να, επιβληθούν κάποιες κυρώσεις, ένας μηχανισμός ο οποίος να λειτουργεί ε, για να λογοδοτήσει μια ΜΑΡ. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε για να ξαναγίνουν ξανά τα ίδια. Ε, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. 30-40 χρόνια, ξανά και ξανά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα για την κοινή γνώμη της Μιαμάρ. Ακούστε, η προπαγάνδα είναι πολύ ισχυρή εκεί. Υπάρχει μια ρητορική μίσους που επικρατεί στη χώρα, αλλά οι νέοι άνθρωποι, όπως είπα και νωρίτερα, ε, είναι αυτοί που μοιράζουν φυλάδια στον κόσμο, στον δρόμο, ε, προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι είναι καλό να αμφισβητηθεί η να, ε, να λογοδοτήσει η Μιαμάρ ε, πρώτων διεθνών δικαστηρίων, αλλά και οι αρχές της Μιαμάρ καταπιέζουν τους ανθρώπους αυτούς Χρειάζονται λοιπόν και αυτή τη βοήθειά σας, τη βοήθειά μας. Χωρίς αυτούς ε, δεν πρόκειται να μπορέσει να αλλάξει η άποψη της κοινή γνώμης. Και γενική... Ε, δεν πρόκειται να αλλάξει και γενικά το τι θα συμβεί στη Μιαμάρ στο μέλλον. Αυτοί είναι μπορούν να αλλάξουν ε, την κοινή γνώμη. Μπορεί να συμβεί, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη απ' έξω, έτσι ώστε το στρατιωτικό καθεστώς, το τυραννικό καθεστώς Μιαμάρ να μην τους αγγίξει. Έγινε λόγος ε, και για τις ανησυχίες που υπάρχουν επί τόπου. Ελπίζω να κατάλαβα καλά το ερώτημα. Εάν ε, δεν έχουμε πρόσβαση στη χώρα, θα είναι πολύ δύσκολο να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Μιλάω υπό το ανθρώπου όπου όλη η οικογένειά μου αυτή τη στιγμή ε, κρατείται, ζουν στο φόβο όλοι αυτοί, δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, ε, δεν κρατούνται, είναι σε κέντρο προσφύγων και υπάρχει αυτή η ρητορική από τις κυβερνήσεις, ε, του στρατό, την αστυνομία, γενικότερα τις αρχές επιβολής του νόμου. Καθώς ε, λαμβάνει η χώρα αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο, τους ρώτησαν ε, τι του συνέβη, πότε υπήρξε αδικία εις βάρος τους, κατά πόσο ε, τους έχουν πάρει ε, περιουσιακά στοιχεία, τα ζώα τους και όταν κάποιοι από αυτούς διαμαρτύρονται τότε τους λένε φέρτε το, το Διεθνές Δικαστήριο ε, αυτή είναι η φίλη σας και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί ε, στο Κοινοβούλιο Όπως είπαν και άλλοι ευρωβουλευτέ, πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Στη χώρα, ιδάλλως, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε κανέναν. Τώρα για το θέμα της ασφαλούς επιστροφής και το κατά πόσο πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν και τα εγκλήματα του παρελθόντος. Εάν δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι από το 2017 υπάρχει μια εικόνα από δορυφόρο που συλλέγει ένα Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής νομίζω στην Αυστραλία έχουν δημιουργηθεί 45 στρατόπεδα, 6 στρατιωτικές βάσεις από το 2017 έτσι έως σήμερα Δεν βλέπω λοιπόν επαναπατρισμό ή επιστροφή σύντομα, τουλάχιστον με αξιοπρεπή και ασφαλή τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νίκολας, ε, θα είσαι ο τελευταίος ε, που θα μιλήσει για δύο λεπτά.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 to resettle, to, to, for the return of those who are refugees back into the country. Thank you. Merci, merci beaucoup, euh, Nicolas. Η πρόεδρος, Νίκολας, σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, πραγματικά, ε, η συζήτηση με τον Νίκολα και τη Γιασμίν. Μισό λεπτό, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, Φιλ. Διακόπτη. Όχι, θέλω να διαφωνήσω ότι δεν αμφέβαλα για την διαδικασία της ποινική δίωξης των ε, τελευταίων των εγκλημάτων. Απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να κοιτάμε και τα δύο θέματα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Φίλοι, σε ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Άρα, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με την ε, μειωμένη, πάμε για τις υπορικές προτιμήσεις, για τον πολιτικό διάλογο και Αύριο πρόκειται να κριθεί από το Διεθνές Δικαστήριο το θέμα της γενοκτονίας. Οπότε θα πρέπει κάτι να κάνει να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Μιανμάρ. Οπότε να περιμένουμε την ε, αυριανή απόφαση και τα όσα πει η Επιτροπή των ε, α, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω ότι βεβαίω ο καθένας εδώ κάνει συζητήσεις του. Ε, Ιζαμπέλ και Ιζαμπέλ, παρακαλώ πάρτε θέσεις. έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αρχίσουμε και να δώσουμε το λόγο όσο γίνεται πιο γρήγορα στους προσκεκλημένους μας Ξέρετε ότι η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισίας ε, είναι... έχει ιστορία, είναι σημαντική και σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο των δικαιωμάτων, σε επίπεδο διακυβέρνηση, σε οικονομικό επίπεδο. Πολλά λοιπόν ζητήματα μπορούν να συζητηθούν. Η κατάσταση στην Ισία σήμερα σε πολιτικό επίπεδο επίσης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μετά τις επαναστάσεις ε, ε, υπάρχουν μια σειρά από διαστάσεις ε, το σύνταγμα τα δικαιώματα των γυναικών που έχουν πραγματικά εξεταστεί σε βάθος μιλήσαμε και για τη Λιβύη και τον αντίκτυπο της αστάθειας στη Λιβύη στις γειτονικές χώρες όπως η Τινησία περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση παρόλα αυτά Πρόκειται για μια κατάσταση που προχωράει, που εξελίσσεται, που σταθεροποιείται. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας ε, ο Καμέλ Τζεντουμπί, ο οποίος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Euromed, πρώην ε, υπουργός των θεσμικών των σχέσεων των θεσμών με την κοινωνία των πολιτών και μαζί μας είναι και η Widet Bouchamaoui η οποία ε, είναι κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2015 και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, της Ισιακή Μηχανίας Εμπορίου και Βιοτεχνίας. Κανονικά πρέπει να δώσω το λόγο και στον Αντρέα Κοτσολίνο, ο οποίο είναι πρόεδρο τη αντιπροσωπεία με το Μαγκρέμπ, που θα την αντικαταστήσει όμω ο κ. Μαγιορίνο, διότι ο κ. Κοτσολίνο ε, ασθενεί δυστυχώ θα δώσω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Μαγιορίνο που το αντικαθιστά και θα πει δύο λόγια στο όνομά του. Bonjour. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την υποχρέωση να αντικαθιστήσω τον συνάδελφο Κατσολίνο που είναι άρρωστος και θα ήθελε πάρα πολύ να παρίσταται. Και ζήτησα να σας διαβάσω ένα σημείωμα από πλευράς του. Εννοείται ότι συμφωνώ με αυτά που διατυπώνει και ευχαριστώ την ε, Μαρία Ρένα διότι κάλεσε την ε, αντιπροσωπεία μας σε αυτή τη σημαντική ε, συνάντηση όσον αφορά την εταιρική σχέση μας με την, ε, την Και τώρα σας διαβάσω το κείμενο Κατσολίνο. αγαπητοί μου, επιτρέψατε πρώτα-πρώτα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Με μεγάλη μας χαρά σήμερα σας φιλοξενούμε ως πάρα πολύ εκλεκτούς εκπροσώπους θεσμών της χώρας σας και έτσι πιστεύουμε ότι θα βοηθηθεί η δημοκρατία σας και οι σχέσεις μας οι κοινωνικονομικές που και έτσι φυσικά αυτό θα έχει επίδραση στο πολιτικό σύστημα από τον Νοέμβριο του 2012 έχετε γίνει ε, εξέχον προνομιούχος ε, εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πλαισιώνει την δημοκρατικό σας μετασχηματισμό του, Ιανουαρίου του 2011 και δεύτερα έχω κάνει κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις ούτω ώστε να παγιωθεί ε, αυτή η μετάβαση και η κοινωνικονομική αλλαγή Πρέπει να έχουμε ορατά αποτελέσματα από αυτή τη συνεργασία και 15 Τρίτου του 18 το Συμβούλιο, το αρμόδιο καθώς τις τι ε, ε, προτεραιότητε τη της συνεργασίας μας 18 με 20 ε, φιλόδοξη συνεργασία κοινωνικονομική ε, βιώσιμη ανάπτυξη, για δημοκρατία, ε, χρηστή διακυβέρνηση, για ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για την ε, γειτονία των χωρών μας, για μετανάστευση, καταπολέμηση τρομοκρατίας κλπ. Και ιδίω εστιαζόμαστε στα θέματα της νεολαίας και αυτό είναι ζήτημα οριζόντιο για όλες τις άλλες πολιτικές. Η Ένωση και η Τινησία έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ζήτημα της συνεργασίας πέραν του 20 και έχουμε τη φιλοδοξία ούτω ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο την προσεγγίσή μας και στο πλαίσιο των ε, διαγνωστικών μας σχέσεων η αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Μαγρέμπα νέκαθεν εστίαζε την δραστηριότητά της στο να βοηθήσει την δημοκρατική αλλαγή, την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα σας και έχουμε παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή τις προεδρικές εκλογές αλλά και τις κοινοβουλευτικές του 19. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την νεαρή σας δημοκρατία. Πρόκειται ε, για παράδειγμα προς ε, μίμηση αυτό το οποίο καταφέρατε εσείς μόνο από όλες τις άλλες εξελίξεις της ε, Αραβικής Άνοιξης βέβαια. Τώρα υπάρχουν διαρροτικά προβλήματα, είναι ευάλωτη η κατάσταση, προβλήματα σε οικονομία, σε συνθήκες διαβίωσης, σε ανεργία που φτάνει στους νέους του 30%. Υπάρχουν ανισότητες μεταξύ παραλίων και εσωτερικού της χώρας και ενδοχώρας και υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα στην γειτονική σας ε, Λιβύη. Επομένως, ε, ακόμα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και βέβαια είναι θετικό το ότι πρόεδρος έχει καταφέρει να βρει την αναγκαία συνένεση, ούτως ώστε να σχηματιστεί σύντομα μια κυβέρνηση και έτσι να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική και η οικονομική μετάβαση και να παίξετε ε, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, να επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα που αμέσως θα έχει και στην οικονομία θετικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και τις ε, επαφές μας με την Διεγνωτική Επιτροπή μας του 2016 για να έχουμε τις επαφές μας αυτές με τους ε, ερετούς σας ε, άρχοντες και εκπροσώπους. Οπότε θα πρέπει να έχουμε την διαβίβαση των καλύτερων εμπειριών για μετανάστευση, ασφάλεια και σωστή διοίκηση και ο κύριο Κοτσολίνη θεωρεί ότι η σημερινή συνάντηση είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι τόσο ώστε να μπορέσουμε να σα ακούσουμε και να μα ακούσετε και να καταλάβουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε. Και εκεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να δούμε ακριβώ εσεί τι ανάπτυξη υποθείτε για τη χώρα σα. Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο για τα όσα είπατε. Και ευθύ αμέσω να δώσουμε τον λόγο ε, στην κυρία Μπουσαμαβή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Με τιμά η παρουσία σας εδώ να σας μιλήσουμε για την χώρα μας, για τους τινήσιους και τις τινήσεις. Όσοι έχετε παρακολουθήσει τη διαδρομή μας, ξέρετε τι έχει γίνει. Ήταν ειρηνική η διαδρομή αυτή, και δημοκρατικέ εκλογές για μας αυτό τον εξαιρετικό χαρακτήρα γεγονό και επίσης υπήρχε και κάτι άλλο το ξεχωριστό η διαφυγή από την ε, δικτατορία προς την ε, δημοκρατία εκεί που να έχουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να αποδεχόμαστε τις διαφορές μας. Πρόκειται για κάτι καινούριο για μας. Ε, Τι μαθαίνουμε τώρα την δημοκρατία. Χρειάζεται χρόνος να έχετε υπομονή. Δεν γίνονται όλα από το βράδυ στο το πρωί. Είμαστε δημοκρατική χώρα, υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ελευθερία τύπου, γίνανε ελεύθερε δημοκρατικές εκλογές και υπήρξε η ελευθερία επιλογής των, των βουλευτών, του Προέδρου. Κάτι το οποίο ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό, σε λίγο χρόνο έγινε και όπως σωστά είπατε ακόμη υπάρχουν ανησυχίε, ε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν θα θέλει η νεολαία μας δουλειά ε, καλύτερη ζωή να μπορούν να εκφραστούν και να είναι ευτυχισμένοι είναι μια πρόκληση το ότι βρισκόμαστε στην αγαπημένη μας ε, περιοχή, την Βόρεια Αφρική, το Μαγκρέμπ, την ε, Μεσόγειο. Δύο βήματα από την Ευρώπη. Και μια χώρα που έχει πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Έχουμε και την ε, γείτονα Λιβύη που έχουμε ιστορικές στενές σχέσεις, αλλά τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική απειλή από την ε, Λιβύη. Η αστάθεια, πάρα πολλά ερωτηματικά, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε ούτως ώστε κάτι να γίνει για αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε τώρα το τι κάνουν άλλοι, τι κάνει η διεθνής ε, κοινότητα και διάφορες χώρες για την κρίση στην Λιβύη αλλά οι πρώτοι που φυστάμαστε τι συνέπειε είμαστε εμείς, τι αρνητικές συνέπειες του εμφυλίου στην ε, Λιβύη. Εμείς, η Τινησία. Ασφάλεια, Πολλέ κυβερνήσεις, προβλήματα οικονομικά, παράλληλο εμπόριο, δεν υπάρχουν άμεσες διμερείς σχέσεις. Και είναι το θέμα του τι πρέπει να κάνουμε, τι υποδομές στα σύνορα και στο εσωτερικό. Όλα αυτά κοστίζουν. Όλοι και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση μας το λένε ξεκάθαρα. Σας βοηθάμε. Εσείς παίρνετε τα περισσότερα, αλλά αυτά είναι σταγόνα το ωκεανό γιατί οι θυσίες μας είναι πολύ μεγάλες, η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Στο επιχειρηματικό έχουμε χάσει πάρα πολλά. Γιατί είχαμε εξαγωγές προς τη Λιβύη, ε, ήταν εύκολες οι μεταφορές, τίποτα τώρα. Όλα τώρα έχουν φρενάρει. Παραεμπόριο, Πάνε και οι δασμοί, ε, πάει, πάνε τα πιστοποιημένα διεθνώς προϊόντα, οπότε και εμείς τώρα χάσαμε και από ρυθμούς ανάπτυξης επίσης η Αλγερία από την άλλη μεριά εκεί υπήρξε ελπίδα δημοκρατίας αλλά ακόμα και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον οπότε και ανησυχούμε Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πλούσια χώρα. Οι περήφανοι που είμαστε μεταξύ αυτών των δύο χωρών δεν έχουμε πρώτες σύλλες, αλλά έχουμε εμπειρία, έχουμε ανθρώπινους πόρους, ε, ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια ως γυναίκα πρέπει να σας πω ότι επίσης είμαστε περήφανες που στον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο είμαστε από πιο προχωρημένους και εκεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Μας ζηλεύουν γι' αυτό πολλές αραβικές χώρες. Χάρη στην ηγεσία του Μπουργκίμπα. Όλα αυτά. Είχε οξυδέργεια και αυτά για το τις σχέσεις μας δηλαδή αλλά επίσης και σε σχέση με το Μαρόκο ε, και οπότε είχαμε δύο πόντους ανάπτυξης που χάθηκαν πολλές οι συνέπειες επομένως σε οικονομικό επίπεδο και όπως είπατε κύριε Μαγερίνο ότι είμαστε σε σωστή ρότα, σε σωστή κατεύθυνση πάμε για την, τον δημοκρατικό μας, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ευάλωτα γιατί πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα σε οικονομικό επίπεδο. Είναι καλά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα στην υγεία και στην ε, εργασία, τα οικονομικά δικαιώματα. Το δικαίωμα του να ζει κανείς ελεύθερος και με ασφάλεια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οπότε και εμεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για τη χώρα μας. Αλλά βέβαια χρειαζόμαστε έναν στρατηγικό εταίρο που πιστεύει στις ικανότητές μας και αυτή η συνεργασία να είναι ωφέλιμη για όλους. Όχι μια μικρή χώρα ε, που κανένας θα πρέπει μόνο να βοηθάει. Ε, να είναι ένας αυθεντικός εταίρος. να συνεργαστούμε για να προοδεύσουμε και να πάει καλά αυτή η συνεργασία και να φέρει ευημερία. Πρόκειται για πρόκληση. Βέβαια, εξαρτάται το πόσο θέλει ο καθένας να πάει καλύτερα αυτή η, εταιρική σχέση. Μια σημαντική νέα εμπειρία, αλλά πολύ ευάλωτοι. Βέβαια χρειαζόμαστε έργα υποδομής, ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε τις πολυεθνικής και τα έργα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια ή να πιστέψουμε ότι είναι η νέα χώρα μας μια χώρα που δεν είναι τόσο ε, πλούσια αλλά που έχει αυτοπεποίθηση για, για το ανθρώπινο κεφάλι, του ανθρώπινους πόρους. Κατάρτιση, εκπαίδευση, υγεία, όλα αυτά που μας δίνουν αυτή την ξεχωριστή θέση στον αραβικό κόσμο, στον κόσμο και στην Ευρώπη. οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε λέγοντας ότι πολλές φορές δείχνουμε κάποια ανυπομονησία. Πολλές φορές υστερούμε χρονικά για τον σχηματισμό κυβέρνηση, για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα τις κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά μας χρειάζεται χρόνος, 9, 10 χρόνια. Μα τι είναι αυτό μέσα στην ιστορία μιας χώρας. Μα χρειάστηκαν εδώ πέρα αιώνες για να φτάσουμε στη δημοκρατία και για να γίνουμε μια ανεπτυγμένη χώρα. Άρα όλα θα γίνουν με συνειδητοποίηση της κοινωνίας, με τη βοήθεια των συνεργαστικών οργανώσεων, με κοινωνικό διάλογο, συνεργασία, συνένεση. Θα τα καταφέρουμε και επίσης ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι τολμηρή. Θα κάνει τις σίγουρα δύσκολες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, όμως θα γίνουν αποδεκτές από το λαό μας. Σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας για τις τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Μπούσα Μαουή. Να δώσουμε τον κόσμο στον κύριο Καμέλ Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση και μάλιστα μαζί με την κυρία Μπούσα Μαουή. βρίσκομαι και πάλι σε αυτό το χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, παραμένει ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στην Τινησία. Ε, χαιρετίζω και την παρουσία της αυτού πρέσβη της ε, Τινησίας. Είναι τιμή για μας που είναι σήμερα παρόν μαζί μας. Όπως είπε και η κυρία Μπουσαμαουή, το περιφερειακό μας πλαίσιο είναι γεμάτο απειλές και σε εθνικό επίπεδο μετά τις εκλογές Χαρακτηρίζεται η χώρα από την περίοδο ε, δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών καταστάσεων μετά τις εκλογές. Χαιρετίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δέσμευσή του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών στην Τινησία. Ίσως κάποιοι από εσά να θυμάστε το πρώτο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Μαΐου του 1996. Πάνε περίπου 25 χρόνια από τότε. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή των συμφωνιών ευρωμεσογειακής συνεργασίας από την Τινησία. Ένα ιστορικό ψήφισμα που επιμένει για το θέμα του αμοιβαίου σεβασμού των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές. Εκείνη την εποχή εξέφραζε την απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλων των ομάδων, πρέπει να τονίσω, όλων των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε, ε, που είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την ε, δίωξη των θυμάτων και των πολιτικών αντιφρονούντων και των οικογενειών τους και εξέφραζαν και την ανησυχία τους για την ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του τύπου κλπ. Έκτοτε η Τινησία έχει κάνει σημαντικές πρόοδους για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την ε, επανάσταση του 2011 κυρίως. Το Σύνταγμα του 2014 ε, σίγουρα εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίω ε, το κεφάλαιο 2 που αφορά τα, τις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε πολλά άλλα άρθρα αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρω το άρθρο 6 για την ελευθερία τη συνείδηση. Και νομίζω ότι είναι η μόνη χώρα στον αραβικό κόσμο που αναγνωρίζεται στο Σύνταγμα η ελευθερία συνείδησης αλλά και σε άλλα σημεία του συντάγματος, το προήμιο παραδείγματο χάρη, Υπάρχουν δεσμεύσεις σαφείς και εγγυήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο για το θέμα της ηθαγένειας. Επικύρωση των διεθνών μέσων για ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, το 2011 το 2017 ψήφισμα κατά της βίας κατά των γυναικών που ετέθησε ισχύ το Φεβρουάριο του 2018 όπου αποτελεί σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο του κινήματος χειραφέτησης των γυναικών στην Τινησία βάσει των ιδεών των μεταρρυθμιστών του 19ου και 20ου αιώνα, Τάρλε Χαντέτ Παντέτ μεταξύ αυτών. Επίσης, ε, ο νόμος ο οποίος ποινικοποιεί την διακριτική μεταχείριση με βάση τη φίλη για μας. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό με βάση την ξεχασμένη μας ε, κληρονομιά που ήμασταν η πρώτη ε, μουσουλμανική χώρα όπου καταργήθηκε η δουλεία το 1846. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που θα ήθελα να αναφέρω εν παρόδο. Μηχανισμοί για την καταπολέμηση των βασανιστήριων, για την πρόσβαση στην ενημέρωση, σχέδια νόμων για, ε, παραδείγματος χάρη, για την ισότητα στα κληρονομικά δικαιώματα, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, και κώδικας που έχει υποβληθεί στην ε, Βουλή για τις ανθρώπινες ελευθερίες. Αυτά είναι διάφορα έργα που πολλές φορές πηγάζουν από καινοτομίες στην Τινησία και πέραν των συνόρων της. Από το 2011 έχουν γίνει πέντε ειρηνικές εκλογές στην Αττινησία και πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις για δίκες πλουραλιστικές εκλογές. Το 2011, το 2014 προεδρικές εκλογές, δημοτικές εκλογές το 2018, ε, βουλευτικές εκλογές το 2019 και η δημοκρατική διαδικασία ε, στην Τινησία δεν ε, έχει ομοιότηση στον αραβικό κόσμο και εντάσσεται στο πλαίσιο των τελευταίων δύο αιώνων στη σύγχρονη Τινησία. Από εδώ ξεκινούν οι στρατηγικές ε, σκέψεις από βασικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Τινησία στο πλαίσιο του διαλόγου που ξεκίνησε από το δίκτυο Euromed από το 2014 μέχρι σήμερα. Αυτή, αυτός ο προβληματισμός και τα αποτελέσματα τα έχετε στην έκθεση που σας δόθηκε, που μιλά για μια εταιρική σχέση της Τινησίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ψηφίσματα και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται, ε, αφορούν τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την κατάσταση εντός της Τινησίας. Μιλάμε για τη δημοκρατική διαδικασία που είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας και της κοινή πολιτικής μνήμης που δημιούργησε ε, την ε, κοινωνική και πολιτική συνένεση για την Επανάσταση. Αυτή η συνένεση υλοποιήθηκε ε, παρά την αυταρχική εξουσία, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, αποδεικνύοντας την δύναμη της τοπικής κοινωνίας παρά τις συνεχιζόμενες ε, δυσκολίες. Και παρότι η κοινωνία των πολιτών δεν είναι πάντοτε ικανοποιημένη από αυτά τα οποία ακολούθησαν. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, όπως ε, πολύ συχνά αναφέρεται πολλοί από εσάς ευρωβουλευτές και πολλοί από τους ηθήνοντες στην Τινησία. Υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις που δημιουργούν ε, σίγουρα και απειλές ε, ε, οι οποίες εντείνονται μάλλον από τις περιφερειακές απειλές. Η Τινησία έχει πολλές προκλήσεις, αλλά βασίζεται στις ίδιες δυνάμεις της, στους ανθρώπους της και θέλει να βασίζεται και στην υποστήριξη που στηρίζεται στην εταιρική σχέση, ιδίω με του γείτονέ τη από την άλλη πλευρά τη Μεσογείου, δηλαδή τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλέ οι προκλήσει, είναι πολλέ οι απειλέ Είμαστε μια μικρή χώρα της Μεσογείου που θέλει να ενταχθεί στη δημοκρατική κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι Τινήσοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιστό στις δεσμεύσεις του και παραμένει πιστό σύμμαχος της Τινησίας στην αναζήτηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και η χώρα μας είναι μια πηγή έμπνευσης και σεβασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Καμέλ Τζεντουμπή για αυτήν την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη μας. Ιζαμπέλ Βίσλερ για το ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Πρέπει να πω ότι παρακολουθούμε έτσι με ικανοποίηση ε, της εξελίξης στην Τινησία ήθελα να θέσω απλά κάποια ερωτήματα για να δω πώς βλέπετε και τη συνέχεια τα προβλήματα που προέρχονται από την τρομοκρατία ε, θεωρείτε αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρότερος κίνδυνος ε, ή εξακολουθεί να είναι εξίσου σημαντικός. Σε σχέση με τη θανατική ποινή, η οποία ε, εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως δεν εφαρμόζεται, αλλά υπάρχει. πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια προοπτική να καταργηθεί και κάτι ακόμα ναι, πραγματικά ε, δεν θέλουμε να δώσουμε μαθήματα έτσι σε καμιά περίπτωση και σε κανέναν. Πώς βλέπετε την κατάσταση με τους πρόσφυγες στη χώρα σας. Και τέλος, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, πώς βλέπετε την ε, εξέλιξη ε, για μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των και γυναικών στην Τινησία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ Ραφαήλ Γκλουξμάν για την ομάδα S&D. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ξέρετε, ε, όλοι βλέπουμε την Τινησία ως μοντέλο δημοκρατικής μετάβασης, ένα μοντέλο δημοκρατίας την οποία οικοδομούν οι ίδιοι την ίση που δεν είναι προϊόν εξαγωγής ε, ε, βομβών και μαχητικών είναι ένα εργαστήριο, αν θέλετε, ένα πείραμα ε, δημοκρατίας ε, για όλη την περιοχή και αν θέλουμε να νικήσουμε ε, τις ε, σκοτεινές δυνάμεις στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο πρέπει πραγματικά να, να στηρίξουμε την δημοκρατία της Τινησίας που είναι ένα αντιπαράδειγμα σε σχέση με αυτά που γίνονται αλλού. Υπάρχει ενίσχυση, υπάρχει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα λοιπόν, πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, από το ζητήμα των επενδύσεων, συγκεκριμένα πολιτικά, ε, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, προ τα που πρέπει να σπρώξουμε τις, τα δικά μας θεσμικά όργανα για να σας βοηθήσουμε και ιδιαίτερα να απευθυνθούμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που είναι το κλειδί για την επιτυχία ε, της ε, εμπειρίας αυτής της θυνησίας. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας χωρίς να παρεμβαίνει όμως μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους νέους ανθρώπους να ε, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να ε, καταρτιστούν και να συμμετάσχουν και στην πολιτική ζωή. Ε, το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με αυτές τις ανταλλαγές. Η πολιτική θεωρήσεων και η δυνατότητα τελικά διέλευση της Μεσογείου. Μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή με την Τινησία, διότι ε, ένα προβλήματα στις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι ότι ε, δεν κάνουμε επαρκή διαχωρισμό μεταξύ των εταίρων μας. Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή μια συμφωνία με το Βιετνάμ, δεν είχα καμία σχέση αυτό βέβαια, ενώ από την άλλη πλευρά της Μεσογείου, εδώ απέναντι υπάρχει μια δημοκρατία που χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί και, και ποια είναι τα συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε για συγκεκριμένη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ ο Phil Binion για τους, για τους Renew. Ναι, δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω. Βεβαίως έχω να κάνω με την οικονομική ανάπτυξη και τα δύο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είχα τη χαρά να επισκεφθούν την Ισία όταν συντάσατε το Σύνταγμα και συνάντησα τότε τον κύριο Γκανούση και άλλους πολλούς ε, ε, και παρακολούθησα με ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια ε, για να δω πόσο ανθεκτική είναι η Ισία μετά την Αραβική Άνοιξη και μετά βεβαίως την κατάρρευση της Αραβικής Άνοιξης αλλού. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν για αυτό που έχετε κάνει ως τώρα που, και που προχωράει τελικά αυτή η δημοκρατική διαδικασία. Τώρα, ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Ε? Ε, μέρη είναι κάτι που συνδέεται με την ασφάλεια, ε, διότι η τουριστική, βιομη, η τουριστική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική και κάθε φορά που υπάρχει κάποια επίθεση, τότε πλήττεται ο τουρισμός στην Τινησία. Ε, ξέρω ότι έχουν, είχαμε πολύ λίγα πράγματα στην επικαιρότητα ε, της Τινησίας. Ε. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε αν υπάρχει κάποια ανάκαμψη σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν πριν από δύο-τρία χρόνια όταν πολλοί τουρίστες εγκατέλειπαν την νησία για λόγους ασφαλείας και μπορούμε να κάνουμε εμεί κάτι για να βοηθήσουμε έτσι ώστε να παραμείνει να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα ασφάλειας ε, και εμπιστοσύνη στην Ισία ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Ε, είπε προηγουμένως ε, η ομιλήτρια, μίλησε για την κατάσταση σχετικά με το εμπόριο στο Μαγκρέμπ διότι είχαμε ένα ψήφισμα κατεπήγον για την Αλγερία πριν από λίγους μήνες και εγώ αναφέρθηκα στην ανάγκη μιας ένωσης του Μαγκρέμπ μετά από μια επίσκεψη στο Μαρόκο τον Νοέμβριο ε, όπου φάνηκε το θέμα αυτό να είναι εξαιρετικά επίκαιρο μιας και τα κλειστά σύνορα με την Αλγερία μου είπαν στο Μαρόκο εντάξει πολύ καλή σχέση με την Ισία πολύ κακές σχέσεις με την Αλγερία όμως ε, και οι κακές σχέσεις με την Αλγερία ε, ουσιαστικά δεν επέτρεπαν την οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο του Μαγκρέμπ ε, ήταν κλειστά τα σύνορα ε, Νομίζω ότι υπήρχε ελπίδα με την πολιτική αλλαγή στην Αλγερία ότι μπορεί να υπήρχε μια νέα προσέγγιση. Ε, στο Twitter ε, έβλεπα παντού μηνύματα αφήστε μας ήσυχους ε, ασχοληθείτε, καθίστε στα αυγά σας αυτά βέβαια από την Αλγερία, από αλγερινούς αξιωματούχους μετά από αυτά που είχα πει στο Κοινοβούλιο. Δεν είμαι λοιπόν τόσο αισιόδοξο όσο ήμουν στην αρχή. Εν πάση περιπτώσει, ε, Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε για να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, στο Μαγκρέμπ ε, και με την Αλγερία για να μπορέσει να επιληθεί αυτό το γεωγραφικό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τον λόγο στη Σελήμ Μαλιμπού εκ μέρους των Πρεσίνων. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω την ερώτηση του γλυξμάντου συναδέλφου Νέα Δημοκρατία ζορίζεται από τους γείτονέ τη αυτό είναι η χώρα σας και οπότε πρέπει να δούμε τι άλλες μορφές δημοκρατίας. Τέτοιες που να δίνουν περισσότερο λόγο στους πολίτες, πιο ενεργό ρόλο. Ε, Βεβαίω και πρόκειται για παράδειγμα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, για νέε μορφέ δημοκρατία. Αυτά τα ζητήματα αναδύονται από όσα είπατε. Επίσης κάτι άλλο. Ε, μία από τις μεγάλες σας προκλήσεις που ε, είναι τι θα γίνει με την οικολογία στα πλαίσια της οικονομικής προσπάθειας, με τα κοινωνικά θέματα, τα εκπαιδευτικά, με τα θέματα υγείας. Και επίσης είπατε, κυρία, ότι θέλετε για αυτήν την δημοκρατική ε, αλλαγή κάποια βοήθεια. Τι είδου βοήθεια θέλετε από πλευρά της Πρόεδρος, και εγώ έχω δύο ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που ακούσαμε. Πολλές φορές, ε, όταν έχουμε κάποιες τέτοιες ε, μεταρρυθμίσεις όπως αυτές της Τινησίας, οι πόλεις ε, και ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γίνεται βέβαια και κάποια θέματα όπως τα γυναικεία δικαιώματα και πολλές φορές όμως δεν είναι τέτοια η στάση της ε, υπαίθρου. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά και από πλευράς επίσης των γυναικών της υπαίθρου. Μιλούμε για αυτή την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Λιβύα. Τι προβλέπετε εκεί. Ε, σήμερα το πρωί μα είπε ο εκπρόσωπος της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι όταν υπάρχει μορική συμφωνία βοηθούνται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά αυτό γίνεται όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, λέω εγώ, και σε σχέση με το περιβάλλον το ίδιο ισχύει. Ε, αυτό επομένως είναι εκ των όνου για την, ε, την Ισία να μας πείτε ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία ούτω ώστε να ωφεληθεί ο κόσμος. Να μην δίνει αυτή η συμφωνία μόνο στην Ευρώπη ε, πλέον έκτημα. Αυτά.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 Ξέρετε, δεν δημιουργήθηκε στην Ισία η τρομοκρατία. Είναι κάτι το οποίο υπέστημεν και εμείς λόγω έλλειψης σταθερότητας. Είναι ένα κύμα το οποίο πλήττει όλο τον κόσμο και δεν βρίσκεται κανεί σε ασφάλεια πουθενά στον κόσμο. Ο κίνδυνο ε, αυτός υπάρχει παντού. Και το είδαμε από τρομοκρατικές δράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη και Αφρική, Ασία, Αμερική. Διεθνές φαινόμενο είναι. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτό είναι το να βελτιώσουμε την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση. Δυστυχώς, εμάς τους Τινήσιους μας πλήττει ιδιαίτερα το ότι αν συμβεί κάτι στην Τινησία, ε, ξαφνικά ε, μοιάζει να είναι η Τινησία η μόνη χώρα στην οποία υπάρχει κίνδυνος. όταν υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση σε κάποια άλλη χώρα, δεν απαγορεύονται οι επισκέψει σε αυτή τη χώρα, ενώ την Τινησία την πλήττουν πιο πολύ οι τρομοκρατικέ επιθέσει και νομίζω ότι θα πρέπει να είστε λιγότερο αυστηροί μαζί μα για να ενθαρρύνετε τον κόσμο να έρχεται στην Τινησία. Τρία εκατομμύρια άτομα ζουν από τον τουρισμό στην την Ισία άμεσα ή έμεσα. Αρκεί μία χώρα στην Ευρώπη να εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για να μην πηγαίνουν οι πολίτες της στην την Ισία, δημιουργείται φαινόμενο ντόμινο και θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες εκτός Ευρώπης. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσπαθήσετε να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την, την Έχουν γίνει πολλά μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Προσπαθούμε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πρόληψη. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις. Και τα ξενοδοχεία και οι κρατικές υπηρεσίες ε, κατανοούν καλύτερα πώς μπορούν να προστατεύσουν ε, και τους τουρίστες. Και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση του τουρισμού, ιδίως Γάλλοι τουρίστες και κάποιοι Βρετανοί έχουν επανέλθει και, και Γερμανοί. Δεν είναι σαν το 2010, πάλι είναι μειωμένο, αλλά υπάρχει κάποια πρόοδο σε σχέση με το 2014 και το 2015 ιδίω. Προσπαθήστε λοιπόν να το βάλετε σε, γενικότερο, σε γενικότερη κλίμακα το πρόβλημα. Δεν πλήττεται μόνο στην Τινησία ο τουρισμός και για μας είναι πρόβλημα. Αν βρείτε κάποιο πρόβλημα, κάποιο, κάποια λύση για το πρόβλημα στη Λιβύη, θα περιοριστούν και για μας οι επιπτώσεις. Αν βρεθεί μια ειρηνική λύση για τη Λιβύη, θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις και για την, την Ισία. Για τους πρόσφυγες θα αφήσω άλλους να απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, το 2011, μετά από αυτά τα οποία έγιναν στη Λιβύη, ανοίξαμε τα σύνορα στην Τινησία. Ανοίξαμε τις πόρτες μας, τα σπίτια μας. 1.200.000 Λίβοι ήρθαν στη χώρα μας και δεν ζητήσαμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Με ανοιχτές αγκάλες τους υποδεχτήκαμε γιατί ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση και χωρίς δεύτερη σκέψη τους υποδεχτήκαμε. Και σήμερα υπάρχουν άλλες χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες, αλλά παίρνουν και πάρα πολλά χρήματα και επιδοτήσεις και ανταλλάγματα γιατί υποδέχονται τους πρόσφυγες. Αν κάνετε λοιπόν τη σύγκριση, θα δείτε ποια είναι η θέση και η νοοτροπία της Τινησίας. Για την ισότητα τώρα ανδρών και γυναικών. Για αυτές ε, τις συμφωνίες για τα δικαιώματα ισότητας ανδρών και γυναικών είμαστε από τις πρώτες χώρες. Είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι. και είμαι υπερήφανη γιατί βλέπω ότι η γυναίκα έχει τη θέση που της αρμόζει, υπάρχει σεβασμός και οι γυναίκες είναι παρούσες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και το νομικό πλαίσιο σίγουρα βοήθησε για να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες σε όλες τις θέσεις. Ακόμη και για τον εκλογικό νόμο, οι καινοτομίες επέτρεψαν στις γυναίκες να συμμετέχουν στο κοινοβούλιο και σε τοπικές ε, αρχές. Υπάρχει πολλή δουλειά βέβαια ακόμη που πρέπει να γίνει και αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρχει ισότητα για τις γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο εφόσον αντιπροσωπεύουμε και το ίμιση του πληθυσμού. Να δώσουμε το λόγο και σε κάποιον άνδρα, λοιπόν, λέει η πρόεδρος. Ναι, ναι. Επανέρχομαι στη συμφωνία ε, συνεργασίας. και ελεύθερων συναλλαγών. Η πρόταση που έκανα εγώ είναι να αλλάξουμε την ονομασία της συμφωνίας αυτής. Θα πρέπει να μιλάμε για μια στρατηγική σχέση με την Τινησία. Μια εταιρική σχέση που θα βοηθήσει και την Τινησία και την Ευρώπη. Θα είναι καλύτερα κατανοητή αυτή η συμφωνία και η έννοια την οποία αντιπροσωπεύει. Είναι μια συμφωνία λοιπόν μεταξύ Ισίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να την εξηγήσετε, γιατί δεν είναι απόλυτα κατανοητή σήμερα. Δεν έχει γίνει σωστά η επικοινωνία, δεν έχουμε εξηγήσει σωστά τι είναι αυτή η συμφωνία και ο κόσμος πιστεύει ότι έρχονται ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κατακτήσουν την Τινησία γιατί είναι το μέγεθός του τέτοιο και η εμπειρία του τέτοια που θα το δικαιολογούσε. Πρέπει, πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε τι θα είναι αυτή η συμφωνία και να το συζητήσετε με τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων και των γεωργών γιατί αυτοί θα συμμετέχουν σε μια τέτοια μελλοντική συμφωνία. Αυτή η διαδικασία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει ελεύθερη ε, κυκλοφορία των ε, ατόμων. Γιατί εγώ ως διευθύντρια μιας εταιρείας ε, υπηρεσιών που συμμετέχω σε ένα διαγωνισμό κάθε φορά πρέπει να ζητάω βίζα. Πού να σας λέω τώρα τι χαρτιά χρειάζονται για να πάρεις μια βίζα. Η γραφειοκρατία είναι ατελείωτη. Δεν υπάρχει λοιπόν ελεύθερη κυκλοφορία, δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Όλα αυτά πλήττουν την Τινησία και τους εργαζομένους. Δεν έχουμε ακόμη εταιρική σχέση. Ο κύριος Τζεντουμπή. Ευχαριστώ, μια και δεν υπάρχει πολύ χρόνο, θα είμαι σύντομο. Όπω θα ξέρετε, ίσω ένα μεγάλο μέρο του προπολογισμού του κράτου σχετίζεται με τα ζητήματα ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για την Ισία. Στο παρελθόν ήταν η παιδεία ε, το, το προπολογισμό. Τώρα είναι η ασφάλεια η εσωτερική ασφάλεια. Χρήματα δηλαδή τα οποία αντί να πάνε στην παιδεία, αντί να πάνε στην ανάπτυξη, πάνε στην ασφάλεια. Βλέπετε το διακύβευμα είναι μεγάλο. Και παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από ό,τι μέχρι τώρα. Είναι πολλές οι θυσίες. Βεβαίως υπάρχει κατάσταση στη Λιβύη που είναι η βασική πηγή εξωτερικής απειλής όμως και στο ιστορικό. Ε, εντάξει, υπάρχει ασφάλεια, κάναμε μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό. Είναι πολύ πιο ασφαλής η χώρα, υπήρξε αντιτρομοκρατικός νόμος που επέτρεψε κάποιες πρόοδους. Υπάρχει και μια συνειδητοποίηση πιο σημαντική του πληθυσμού του, της, της τρομοκρατικής απειλής και οι δυνάμεις ασφαλείας προσαρμόστηκαν στην κατάσταση και βεβαίω την αντιμετώπισαν με μεγαλύτερε δυνατότητε. Η συνεργασία ήταν πολύ πιο χρήσιμη με τι ευρωπαϊκέ χώρε στο θέμα αυτό, στο θέμα τη ε, ασφάλεια. Όμω γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λύση τη ασφάλεια δεν αρκεί αν θέλει κάποιο να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία βιώσιμα. Υπάρχουν άλλοι πόροι, ε, οικονομικοί, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν λόγοι ανισοτήτων, άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι. Ε, παίζουν ρόλο όλα αυτά για την τρομοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση, την οποία σιγά σιγά τη δημιουργούμε στην Τινησία, να λάβουμε υπόψη δηλαδή τις αιτίες της τρομοκρατία, τις περίπλοκες αυτές αιτίε, εσωτερικέ, εξωτερικέ, εμεί πάντα θέλαμε να συνεργαστούμε με τις ευρωπαϊκές χώρες για τα ζητήματα αυτά. Βεβαίω ε, υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι σημαντικά. Υπάρχει το θέμα τη θανατική ποινή που σχετίζεται και αυτό με την τρομοκρατία. Εμεί θέλουμε να την καταργήσουμε πρέπει να γίνει μια συζήτηση όμως ε, εθνική στη χώρα. Ε, η θανατική ποινή είναι ντροπή για μας. Το λέω ως υπερασπιστάς δικαιωμάτων. Είναι ντροπή για μια νέα δημοκρατία. Όμως ε, κάποια θέματα πρέπει κανείς να τα συζητήσει. Πρέπει να τα προετοιμάσει, πρέπει να οριμάσουν. Ε, υπάρχουν και κενά. Δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα νόμο για το άσυλο, ένα νόμο που να προστατεύει τους πρόσφυγες. Ε, έχουμε πάρει πρωτοβουλία στου κοινωνικού πολιτών για να προτείνουμε ένα σχέδιο νόμου. Γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο αρχών υπάρχει ήδη ένα σχέδιο στην προπαρασκευαστικό στάδιο. Θα φροντίσουμε λοιπόν αυτό ο νόμο που θα έχει να κάνει με την προστασία των προσφύγων να προστατεύει σύμφωνα με ε, τους διεθνείς, ε, τα διεθνή πρότυπα. Είναι και αυτή μια από τι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κάτι άλλο. Ναι, βεβαίω, ένα από τα διακυβεύματα είναι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σε όλε τι διαστάσει του. Έχουμε μια νεολαία καταρχήν η οποία είναι εκπαιδευμένη. Μεταξύ των εκπαιδευμένων αυτών είναι πολλοί που έχουν διπλώματα αλλά δεν έχουν δουλειά. Για πολλού και διάφορου λόγου. Πάνω από 150.000 άνεργοι με δίπλωμα ε, στη χώρα μου. Υπάρχουν και πολλοί νέοι όμω από την Ήπεθρο, από το ιστορικό τη χώρα. Υπάρχουν κάποια σχέδια ευρωπαϊκά προς την κατεύθυνση αυτή αλλά δεν αρκούν. Είναι πολύ περιορισμένα, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε συνεργασία με την Ισία. Τώρα, οι ανταλλαγέ. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να καταρτιστούν στα πανεπιστήμια, να εκπαιδευτούν στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, στου θεσμού του ευρωπαϊκού, σε διάφορα προγράμματα που έχει δημιουργήσει η Ευρώπη για να βοηθήσει άλλε χώρε τη Ένωση. Α είναι ανοιχτά αυτά τα προγράμματα και για του δικού μα νέου. Έχει γίνει μια αρχή, αλλά πρέπει να πάμε πιο μακριά. Από την άλλη, ε, στην Τινησία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς, δεν, δεν κατέχουμε επαρκώς αυτά τα προγράμματα, αυτές, αυτή την προσφορά που υπάρχει από την ευρωπαϊκή πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε έτσι ώστε ε, να είναι πιο αποδοτικά όλα αυτά και για μας. Το θέμα των θεωρήσεων ε, έχει να κάνει και με μια πτυχή που είναι κάπως παράδοξη, έτσι. Αφενός η Αλέκα θέλει να αναπτύξει μια σειρά από ε, σχέσεις, από ε, συναλλαγές, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν ε, ε, περιορισμοί. Λέμε ελευθερία επενδύσεων, αλλά δεν μπορούν οι επιχειρηματίες να, να μεταβούν και να επενδύσουν στην Ευρώπη. Ενώ οι Ευρωπαίοι μπορούν να έρθουν στην Ισία. Λοιπόν, αντί να αποσυνδέουμε το θέμα του εμπορικού από το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση, σφαιρική. Τα φυτοκοινωνικά κριτήρια έχουν να κάνουν με το ζήτημα του δικαιώματο ε, στην υγεία, ε, το δικαίωμα το περιβαλλοντικά. Όλα αυτά σχετίζονται και με τη γεωργία. Ε, δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε κατακαιρματισμένα. Πρέπει οι διαπραγματεύσεις να είναι σφαιρικές. Τι μπορεί να προσφέρουν βεβαίως οι εμπορικές συμφωνίες στην ανάπτυξη. Και βεβαίω πάντα λαμβάνοντα υπόψη και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Όμω, αν μια εμπορική συμφωνία ε, δεν ενθαρρύνει την Τινησία να επενδύσει περισσότερα στο ιστορικό τη χώρα, στην ενδοχώρα, στην πηγή πολλών προβλημάτων, προβλημάτων που έχουν να κάνουν και με την πολιτική αστάθεια. Ε, αυτό μα δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι Τινησιακέ αρχέ, όλε οι ζωντανέ δυνάμει της χώρα, είναι έτοιμε να συζητήσουν τι ανταλλαγέ με του Ευρωπαίου. Θέλουμε ανταλλαγέ με του Ευρωπαίου αλλά θέλουμε οι ανταλλαγέ αυτέ να λαμβάνουν υπόψη μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Με βάση και τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώς. Η οικολογία ε, δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη από τους διάφορους παράγοντες της νησίας και λυπάμαι γι' αυτό. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή υπέρ μιας ε, παραγωγικής έτσι, ε, Υπάρχει όμως ακτιβισμός ε, στην κοινωνία των πολιτών όλο και πιο συχνά. Πολλοί ηθήνοντες και πολιτικοί ηθήνοντες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να ξαναδούμε αυτήν την σχέση μας με τη φύση, με το μοντέλο που αναπτύσσουμε σήμερα ε, για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Υπάρχει μια συνειδητοποίηση και στις επιχειρήσεις. Ε, δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη, αλλά πρέπει, πρέπει να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Τώρα, πώς μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Ε, πώς η πρόοδος που έχει γίνει αποδεκτή σε έναν βαθμό στις πόλεις θα γίνει αποδεκτή και στην Ήπεθρο. Εδώ ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ενώσεις ε, πολιτών παντού στην νησία και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Αυτές τις ενώσεις, αυτές, αυτές τις οργανώσεις πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο απολογισμός είναι έτσι ε, μέτριος, διότι ήταν, είναι μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, μια θεσμική προσέγγιση. Ε, και εδώ τίθεται το θέμα της σκέψη γύρω μια, μια νέα μορφή δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί μέρος μια ευρύτερη συζήτηση, όχι μόνο στην Τινησία. Οι εκλογές ε, στην Τινησία ε, εξέλιξαν έναν πρόεδρο που θέλει να αλλάξει η πυραμίδα. Αντί να σκεφτόμαστε από πάνω προ τα κάτω, θέλει να σκεφτόμαστε από κάτω προ τα πάνω. Αυτό λέει ο πρόεδρό μα. Γίνεται αυτό. Ε, είναι εφικτό. Είναι μέρο τη συζήτηση. Πολύ την ίση ενδεχομένω ε, να μην είναι τόσο αισιόδοξοι σχέση με αυτή την προσέγγιση και τίθενται πολλά ερωτηματικά. είναι και αυτό μέρο των συζητήσεων για τα όρια τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία σήμερα να λάβουμε υπόψη ε, πραγματικά το τι θέλουν οι άνθρωποι, ποιε είναι οι προσδοκίε του. Δεν θέλουμε βέβαια να αρνηθούμε, ε, να απαρνηθούμε το κοινοβουλευτισμό, την ύπαρξη πολιτικών κομμάτων, την ύπαρξη κοινωνία των πολιτών. Αλλά είναι αυτό και αυτό μέρο τη συζήτηση, μια συζήτηση που, παραλαμβάνω, πάει πολύ πέρα από την Τινησία. Εμεί συμμετέχουμε και νομίζω ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο τα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Συγγνώμη. Ε, η εταιρική σχέση με την Ευρώπη λοιπόν είναι σημαντική και το Ευρωκοινοβούλιο είναι σημαντικό για μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, θεσμοί, μηχανισμοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπλοκοι. Ε, είναι 27 κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν άλλες άλλε ανησυχίε, άλλε προτεραιότητε. Υπάρχει όμω ένα αλλά εδώ. Ε, μην ξεχνάμε ότι έχει σύνορα και με τον Νότο η Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο, ε, την Αφρική. Δεν μπορεί να τα αγνοεί αυτά η Ευρώπη. Δεν μπορεί να μην τα αντιμετωπίσει ισότιμα. Αυτή είναι η έκκληση που θέλουμε εμείς να κάνουμε και θέλουμε να ακουστεί. Και βεβαίως έχουμε και φίλους εδώ στην Ευρώπη, το ξέρουμε. Έχουμε φίλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φίλου τη Δημοκρατία της, της, της δημοκρατίας της Τινησίας. Συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα δώσω το λόγο πολύ γρήγορα για ένα λεπτό στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για να, γιατί έχουμε και την επόμενη συζήτηση. Ευθύς εξ αρχής πάντως να ευχαριστήσω τους προσκεκλισμένους μας από την Τινησία και όλους όσους σήμερα συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Το θετικό μήνυμα που δίνουμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μια δημοκρατία όπως αυτή της Ισία στον αραβικό κόσμο. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Συμφωνούμε με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Συμφωνούμε και με τους βουλευτές και με τους την ισχύουσα εκπροσώπους. Απλώς θα θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις από πλευράς μας να σας πούμε. Είναι εταίρος κλειδί στο Μαγρέμπ για μας. Την έχουμε πλησιώσει σε όλες τις προσπάθειες παγίωσης της νεαρής δημοκρατίας και της προσπάθειας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Επί δεκαετίες και έχουμε πρόθεση να αρχίσει το νωρίτερο δυνατόν η συνεργασία με νέα κυβέρνηση και νέο πρόεδρο. Να υποστρίξουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις και σε αυτά τα πλαίσια ελπίζουμε όπως και ο λαός ότι η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης να ολοκληρωθεί το συντομότερο και βέβαια υπάρχουν πολλέ προκλήσεις, πολλά προβλήματα, θα πρέπει και οι προσπάθειες να ενταθούν. Έχω σας πω τρία παραδείγματα. Έχουμε τις εκλογές του 19, ε, είχαμε φυσικά χρονική πίεση. Εμείς πάντως στείλαμε κάποια εκλογική αποστολή, είναι τώρα στο Τίνιδα, γίνεται αυτή η έκθεση και κατέβηκαν ε, λίγες γυναίκες στον πολιτικό στίβο. Επίσης είχαμε ε, θεσμικές ε, μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει ακόμα να ολοκληρωθούν. Επίσης είναι και το ζήτημα της συγκρότησης του συνταγματικού δικαστηρίου και επισης επίγουν επήγουν κάποιες μεταρρυθμίσεις κοινωνικο-οικονομικές. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές, ιδίω όσον αφορά την περιφερειακή συνοχή και τις ευκαιρίες προς τους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνούμε ότι είναι πρόβλημα ε, η επικοινωνία σε σχέση με τη Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου. Θα πρέπει οι εταίροι μας να μας βοηθήσουν να σταματήσει η κακή εικόνα που έχει η Συμφωνία. Οπότε με την ευκαιρία που έχουμε εδώ τους ταινιουσίους εκπροσώπους, ναι, η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ και επαναλαμβάνω Να μην λέμε ότι είναι το πρόβλημα μόνο επικοινωνία στο πρόβλημα των εμπορικών συμφωνιών. Θα πρέπει να εμπλαγεί η κοινωνία, ο κόσμο και όπως είπατε και εσείς, ε, ως προς το ότι όλοι να βγαίνουν κερδισμένοι και να μην είναι μονόπλευρο το όφελος από αυτές τις συμφωνίες. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει κάπως η ευρωπαϊκή ρητορική σε σχέση με αυτό. Ε, ευχαριστούμε όσα μας είπατε. Και τώρα...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 Euh, και ευθύ αμέσω, λέει πρόεδρο, συνεχίζουμε με την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τα ανθρωπινά δικαιώματα στην χώρα. Βεβαίω και υπάρχουν ε, κάποιοι εδώ που ενδιαφέρονται για το Μαγρέμπ, άλλοι όμως ενδιαφέρονται για την ε, Λατινική Αμερική. Οπότε παρακαλώ ποιοι θέλουν να αποχωρήσουν ή να μπουν, αλλά ήσυχα. Τώρα έχουμε τον ε, Κλάουδιο Νάς από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο. Ε, είναι πανεπιστημιακό σε σχέση με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έτσι θα μπορέσουμε από την χιλή να ακούσουμε πώς έχει η κατάσταση και στη συνέχεια θα έχει το λόγο η κυρία Πατρίθια Πάργα Βέγα. Και συνεχιστεί η συζήτηση. 10 10 λεπτά είπατε και σας δίνουμε το λόγο. Muchas gracias. Ευχαριστώ. πολύ. Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε μια από τις ε, διαδικασίες ε, κινητοποίησης των πολιτών ε, από τις πιο βαθιές στην πρόσφατη ιστορία της Χιλής. Η απάντηση της κυβέρνησης Πολιτικά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 es que a la fecha just one, hay más. Claudio, just, just one minute. Um, uh, Αυτό μισό λεπτό λέει πρόεδρος. Δεν γίνεται διερμηνία. Δεν υπάρχει μετάφραση από το πρωτότυπο τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ακούμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακούγεται η διερμηνία. Μήπως μπορούν οι διερμηνείς να λάβουν υπόψη ότι είναι ο ήχος ε, καλώς. Γίνεται να έχουμε διερμηνία από τα ισπανικά προς τις άλλες γλώσσες. Εντάξει. Some are saying yes and some are saying no. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Problem of hearing. Έχετε πρόβλημα με τον ήχο. Έχετε το κείμενο. Is it possible to have a translation yes or not? Γίνεται να μεταφράσετε ναι ή ου. Γιατί λένε άλλοι ναι και άλλοι όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι λένε ναι και άλλοι λένε όχι. Αν είναι καλός ο ήχος, είναι καλός για όλους. την Donc, je sais pas, moi, je sur la qualité de Δεν ξέρω τι κάνουμε τώρα συμβούλιο σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Αν θέλετε κάντε το, αλλά κάποια στιγμή αυτά όλα μας δυσκολεύουν. Εγώ πάνω από όλου σέβομαι τα δικαιώματα των διερμηνίων, αλλά γιατί λένε άλλοι ναι και άλλοι όχι. Ακούτε ή όχι.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 αλλά θα είμαι αυστηρότερη στο εξή όσον αφορά την διερμηνία. Στα ισπανικά λοιπόν. Okay, uh, sorry, uh, Claudio, you can... Uh, Claudio, λέει ο πρόεδρος, μπορείς να συνεχίσεις στα ισπανικά. Μπορούμε να σε καταλάβουμε. Okay,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 Eh, eh, Ευχαριστώ. Σας δίνω ευθύς αμέσως τον λόγο, Πατρίθια. Έχετε πέντε λεπτά. Ενδεχομένως να έχουμε και την ευκαιρία να έχουμε και μια συζήτηση. Θα στήσω από ε, τους μη Ισπανόφωνους να πάρουν τον λόγο πρώτη, έτσι ώστε να υπάρξει διερμηνία. Πατρίθια, έχετε τον λόγο. Έχετε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής, η απόφαση της κυβέρνησης της Χιλής του κυρίου Πινέιρα να κηρύξει και κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19 Οκτωβρίου 2019 δημιούργησε μεγάλη ανησυχία ε, μεταξύ των, των κοινοτήτων των χιλιανών που ζουν στο εξωτερικό. Τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει να βγάλει το, το στρατό στο δρόμο, ανοίγει μια πληγή η οποία δεν έχει ποτέ κλείσει στη χώρα μας διότι για πολλούς από εμά είναι σαν να ξαναζούμε την ε, ε, δικτατορία του Πινοσέτ. Χάρη στις νέες τεχνολογίες, ε, μια ομάδα συμπατριωτών μας που ζουν στη Βαρκελόνη ξεκίνησαν μια έκκληση έτσι ώστε όλοι οι χιλιανοί οι οποίοι ευαισθητοποιούνται γύρω από το ζήτημα αυτό να μπορέσουν κάπως να εκφραστούν. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 18 ε, Οκτώβρη. Χίλι ξύπνα λέγεται. Ε, ε, η συλλογικότητα αυτή. Ε, δεν έχει σταματήσει έκτοτε όμω η καταστολή. Η καταστολή μάλιστα έχει αυξηθεί, όπως είπε και ο Κλάουντιο Νάς νωρίτερα, ο Δόκτωρ Νάς. Οι διεθνείς οργανισμοί υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκδώσει εκθέσεις και είναι κατηγορηματικές αυτές οι εκθέσεις η Επιτροπή μας έκανε και μια δεύτερη νομική έκθεση με επικαιροποίηση των διαφορών ε, υποθέσεων και να ανακφράσουμε την ανησυχία μας απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Αυτή η έκθεση αναφέρεται σε επίσημα στοιχεία τα οποία αναγνωρίζει ένα ε, ένα κρατικό φορέα, το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γνωρίζουμε βεβαίω ότι οι αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι, διότι είμαστε και σε άμεση επαφή με τι οργανώσει υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χιλή. Οι πολιτικέ επιπτώσει ε, για του. Ε, φοιτητές οι οποίοι θεωρούνται ότι δημιουργούν ε, έκτροπα είναι πραγματικά απίστευτα. Μιλάμε για μαθητές, ανήλικους, οι οποίοι απλά ασκούν το δικαίωμά τους ε, για ανυπακοή. Μιλάμε για ανήλικους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν στο, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιό τους μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι φοιτητικών οργανώσεων, ο Δελγάδο, ο Βίκτορ Σάφρο, η Γερουσία ε, ενέκρινε ένα σχέδιο της κυβέρνησης που δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό ε, να χρησιμοποιεί τη, τις, τις στρατιωτικές δυνάμεις να εξασφαλίσει τις κρίσιμες υποδομές, να διαφλέξει τις κρίσιμες υποδομές. Τι σημαίνει όμως κρίσιμες, υποδομέ υποδομές στην Χιλή. Στις περισσότερες χώρες μιλάμε για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας, νερό, ηλεκτρικό, ε, επικοινωνίες και βεβαίως και είναι σημαντικό όταν υπάρχει άμεση ανάγκη η έκτακτη ανάγκη. Στη Χιλή όμως ε, εδώ όλα αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία είναι στα χέρια ιδιωτών. Είναι στα χέρια του ιδιωτικού τομέα και πάει πέρα από αυτό το project. Μιας και ο, ο πρόεδρος Δημοκρατίας μπορεί μέσω διατάγματος να αποφασίσει ο ίδιος ποιε είναι αυτές οι υποδομές ε, οι, ε, οι κρίσιμες. Είναι πραγματικά παράδειγμα που συμβαίνει στη Χιλή για οποιοδήποτε πολιτικό καθεστώς το οποίο θέλει να ονομάζεται δημοκρατικό. Και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις χώρες που εκπροσωπείτε εσείς εδώ σε αυτό το θεσμικό όργανο. Ε, είναι μεγάλη σιωπή πέρα από κάποιες ε, εξαιρέσεις για αυτά που συνέβησαν στη Χιλή τελευταίες τρεις μήνες και αυτό είναι ντροπιαστικό. Η Χιλή ήταν η πρώτη χώρα της Αναλλακής Αμερικής που, που υπέγραψε συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει επικυρωθεί, που ισχύει η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που προβλέπεται στι διεθνεί ε, αυτέ συμφωνίε, από ό,τι φαίνεται, μένει κενό γράμμα. Τι νόημα έχει να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα, να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα που δημιουργήθηκε ακριβώ για να εφαρμόζεται ε, σε μια περίπτωση όπω αυτή ε, και εφόσον δεν, είναι υποχρεωμένε οι, οι, πλευρέ να το σεβαστούν. Δεν είναι μόνο ευθύνη τη κυβέρνηση, είναι ευθύνη και τη διεθνού κοινότητα που ε, σιωπά και έτσι είναι συνένοχη. Αφού μπόρεσε η κοινωνία η ίδια να ξυπνήσει απέναντι σε αυτές τις καταχρήσεις. Εμείς, το, δίκτυο, Διεθνές Δίκτυο Χιλιανών, ε, σας καλούμε να ξυπνήσετε, να ξυπνήσετε τα θεσμικά σας όργανα για να καταδικαστούν αυτές οι συστηματικές, μαζικές, σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα από το κράτος της Χιλής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πατρίσια. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ισαμπέλ, η οποία μπορεί να μιλήσει πορτογαλικά ε, και στον Φιλ, εφόσον ε, το θέλει για να μιλήσει στα αγγλικά και στη συνέχεια θα το λόγο και στον Μιγγέλ και στον κύριο Αλβάρη που μιλούν και οι δύο ισπανικά. Ισαμπέλ στα πορτογαλικά παρακαλώ. Μπορώ να προσπαθήσω να μιλήσω και ισπανικά. Υπάρχει διερμηνία. Ναι. Μέχρι και μισή. Πρώτα πρώτα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. για να μας πείτε τι για τις εξελίξεις στην χώρα σας. Να σας τα πω πορτογαλικά μια που τώρα έχουμε διερμηνία. Άκουσα μεγάλη προσοχή αυτές τις ανησυχίες σας για τα προβλήματα, την ενημέρωση την οποία μας προσφέρατε και το ερώτημα που προγύπτει είναι πώς κανείς μπορεί να ξεπεράσει αυτή την ε, κρίση. Μπορεί να βοηθούν κάποιες συνταγματικές αλλαγές. Βέβαια η αναθεώρηση του συντάγματος από μόνη της δεν θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα που οδήγησαν ε, σε αυτή την σύγκρουση. Αυτά τα προβλήματα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, πόσοι δυσκολίες θα ξεπεραστούν. Και στα αγγλικά μπορώ να σας ακούσω. Πώς επομένω έλεγα, λέει ο Μιλήτρια, μπορούμε και να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση τη χώρα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να μου πείτε είναι ποιες είναι η, πώς είναι η κατάσταση σχέση με το κίνημα ή τα κίνηματα ε, και τι σχέσεις έχουν τα διάφορα κινήματα με το καθεστώς, με τα θεσμικά όργανα της χώρας. Μόνο με τον διάλογο μπορείτε να βρείτε την διέξοδο. Φιλ, έχεις δύο λεπτά γιατί θα σταματήσει η διερμηνία. Θα ήθελα να μου πείτε εάν τα πολιτικά κόμματα στηρίζουν αυτή την ε, προσπάθεια, αυτή τη διαδικασία Είπατε για δημοψήφισμα, για το αν θα γίνει η δημοτική αναθεώρηση. Συμφωνούν τα πολιτικά κόμματα. Όλα. Ή υπάρχει κίνδυνος αντιρρήσεων για αυτήν την προσέγγιση. Και έχει υπάρξει κάποια ύφεση ή συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες. Έτσι βοηθήθηκε η κατάσταση στο να ε, χαλαρώσει. Κύριε Άλβαρτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω τον Κλάουδιο Νάσου. Στις 18 Οκτωβρίου ξεκίνησε αυτό το κύμα διαμαρτυριών στην ε, χώρα. Περισσότερες ήταν ε, ε, ειρηνικές στην αρχή και κατήγγυλαν τις ανισότητες. Κατόπιν όμως άρχισε ένα κύμα βίας, επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση, καταστροφές σε καταστήματα και έχουμε κάποια στοιχεία. Μιλούμε για δύο δις δολάριο. Οπότε τότε η κυβέρνηση κήρυξε την κατάσταση εκτεκτή ανάγκης. Μετά είχαμε την καταγγελία για κατάχρηση εξουσίας και άσκηση βίας από την ε, ε, αστυνομία. Οπότε ο ΙΕ έστειλε την ε, εκπρόσωπό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να εξετάσει τα πράγματα. Και τον Δεκέμβριο πρόκειψε μια έκθεση και έχουμε όμως και μαρτυρίες και αναφορές και εκθέσεις του Human Rights Watch και είπαν ότι υπήρξε υπερβολική καταχρηστική χρήση βίας αλλά και κάποιον μη επικίνδυνο για τη ζωή όπλων από την αστυνομία. Οπότε υπάρχει τώρα συντονισμός ε, μεταξύ κυβερνητικών αρχών και δικαιοσύνης για να ερευνηθεί η κατάσταση και να υπάρξουν κυρώσεις για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, Τώρα η εισαγγελία εξετάζει το ζήτημα της καταχρηστικής άχρησης ε, βίας και ενδεχομένης παραγωγή στη δικαιοσύνη αστυνομικών ε, και εφαρμόζεται τα σχετικά πρωτόκολλα για χρήση βίας από την αστυνομία και χρήση μη θανατηφόρων όπλων. Ε, οπότε, επίσης, πρόκειται να βοηθηθούν και ενισχυθούν όσοι θύματα της βίας. Νομικά, ιατρικά, ψυχολογικά. Εκείνοι, εκείνοι που υπέστησαν την ε, κατάχρηση εξουσίας. Πασχίζει τώρα η χώρα να υλοποιήσει τις προτάσεις, τις συστάσεις του ΟΗΕ αλλά και του Human Rights Watch αλλά και η Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έχουν καταγραφεί παραδιάστημα δικαιωμάτων από ε, την Εθνική και Ανεξάρτητη Αρχή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επίσης, συνεργασία με δημοσιογράφους και ακτιβιστές, ε, συνεργασία ήταν ε, για τη διερεύνηση των πραγμάτων. Βεβαίω υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση Πινέιρα έχει υλοποιήσει κάποια μέτρα όπως προβλέπει το Σύνταγμα για τις εγγύησεις υπέρ των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά και να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, θα πρέπει να βοηθήσουμε το ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή και να συνεχίσει να κυριαρχεί η ελευθερία στη χώρα. Ευχαριστούμε, Μιγγέλη, Πρόεδρος. Συγγνώμη, δίνει το λόγο στον Μιγγέλη, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους δύο καλεσμένους μας που ήρθαν να μας εξηγήσουν τι γίνεται. Πρώτα πρώτα να καταδικάσουμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγινε στην Χιλή κατά τους τελευταίους μήνες. Αυτό έγινε συστηματικά. Ε, γίναμε μάρτυρες μιας έκρηξης, ε, μιας δυσαρέσκειας κατά του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό δεν έγινε μόνο στη Χιλή, έγινε και αλλού. Και η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η συστηματική καταστολή του λαϊκού κινήματος. Πολύ σημαντικό. Το λένε όλες οι εκθέσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Δεν πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα. Πρόκειται για μια πολιτική, ε, πρόκειται για απόφαση κυβέρνησης και αστυνομίας. Αυτό του είδους η δυσανάλογη καταστολή ε, κληροδότημα της δικτατορίας Πινοσέτ. Δεν έγινε η διαφορά, δεν έγινε ο μετασχηματισμός, δημοκρατική μετάβαση. Ακριβώς όπως φάνηκε αυτούς τους τελευταίους μήνες, γιατί πριν είχαμε βία, είχαμε καταστολή στην Χιλή και φούσκωσε το λαϊκό κίνημα και φούσκωσε και η καταστολή και είχαμε ακριβώς ε, κόσμο που δολοφονήθηκε για, επειδή διαμαρτυρόταν ε, και θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος ε, να γίνουν απρόσκοπτα αυτές οι διαδηλώσεις. Οπότε αυτό καταγγέλουμε την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα του μετρό, δεν είναι πρόβλημα ε, οικονομικό. Πρόκειται για τον ελευθερισμό που έφεραν το άνοιγμα του, του, του, χάσματος ε, μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Γιατί δεν έγινε ο σχηματισμός από την δικτατορία. Οι δικτατορίες κληροδότησαν στην κυβέρνηση αυτές τις πολιτικές που μεγάλωσαν τις ανισότητες. Τελειώνω με, την ερώτηση έχουμε τη συμφωνία. Α, τι να κάνει το κοινοβούλιο, τι μέτρα, πώς να βοηθήσει το κοινοβούλιο και η υποεπιτροπή μας τι να κάνει για να βοηθήσει τον διάλογο και την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στα ισπανικά. Οι διερμηνείς σας χαιρετούν. Claudio, you have the floor. Muchas gracias. Voy